Bien, chers collègues, euh, mesdames et messieurs, bonjour. Veuillez prendre euh, place, s'il vous plaît. Euh. Λοιπόν, καθίστε παρακαλώ. Ο κύριος Ρόντους, ο οποίος θα πρέπει να πάρει το λόγο, θα έρθει σε λίγα λεπτά. Επιστρέφει από το κέρας της Αφρικής σήμερα και κάνει ό,τι μπορεί για να είναι ανάμεσά μας σήμερα. Σε πολύ λίγη ώρα λοιπόν θα είναι εδώ. Αν δεν έχετε άλλες παρατηρήσεις σχετικά με τα πρακτικά, πέμπτη, της 5ης Ιανουαρίου θεωρούνται δεκτά μέχρι το τέλος της συνεδρίασης. Θυμίζω ότι σήμερα το απόγευμα αποκινούμε την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Θα έχουμε μια συνεδρίαση με την κυρία Άστον στην Ολομέλεια θα έχουμε μια ανταλλαγή απόψεων για τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής και της πολιτικής ασφαλείας. Και θα ήθελα, περιμένω να έρθουν και οι υπόλοιποι συνάδελφοι, γνωρίζετε ότι τελευταίες δέκα μέρες στη Γαλλία χαρακτηρίζονται από τραγικά συμβάντα η δολοφονία επτά προσώπων τριών στρατιωτικών και τεσσάρων μελών της εβραϊκής κοινότητας της Τολούζης. Ένα φρικτό έγκλημα το οποίο χτες μάλιστα προκάλεσε θύματα στα παιδιά. Θα ήθελα λοιπόν να κρατήσουμε ενός λεπτού σιγή τιμώντας τα επτά αυτά θύματα εφόσον ε, συμφωνείτε. Euh, Σας ευχαριστώ πολύ. Περιμένοντας τον κύριο Ρόντο, θα ήθελα να κάνω μια εισαγωγή στη σημερινή συνεδρίαση που ασχολείται με ένα θέμα το οποίο έχει αρχίσει, θα έλεγα, να είναι το κεντρικό σημείο της ε, κοινή πολιτικής στον τομέα της ασφαλείας, το κέρας της Αφρικής ουσιαστικά. Έχουμε πολλές δραστηριότητες εκεί Έχουμε την επιχείρηση Αταλάντα η οποία ξεκίνησε μετά το τέλος του 2008. Η επιτυχία της έχει καθολικά αναγνωριστεί. Πρόκειται για μια αποστολή η οποία έχει περάσει από πολλές εξελίξεις με διαφορετικούς τρόπους λειτουργίας και εξάπλωσης πιο περίπλοκους από ότι στην αρχή της λειτουργίας της με πιθανές ε, εξαπλώσεις της δραστηριότητας αυτής ε, ε, σε, σε υπηρετικά πλέον εδάφη και τη συμμετοχή επίσης ενόπλων στρατιωτών στα σκάφη τα οποία κάνουν τις διοψίες. Υποδεχόμαστε σήμερα λοιπόν τον Αβαρχοπότς, ο οποίος ε, είναι υπεύθυνο ε, για την επιχείρηση αυτή, είναι ο αρχηγός της επιχείρησης αυτής από το στρατηγείο της Μεγάλης Βρετανίας. Ξέρετε ότι υπάρχει και μια αντιπροσωπεία της δικής μας επιτροπής, η οποία είχε επισκεφθεί ε, την περιοχή. Πέρυσι την προηγούμενη εβδομάδα στην Ολομέλεια του Στρασβούργου έγινε και μια συζήτηση για την ναυτική πειρατεία. Είναι ένα θέμα πάνω στο οποίο, εν πάση περιπτώσει, είναι πρωτοπόρος η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέλει να ασκήσει πλήρως τις αρμοδιότητες του, έτσι ώστε να συμπληρώσει αυτή τη σημαντική δραστηριότητα με τον κύριο Ρόντο, τον οποίο είχαμε υποδεχθεί και στο τέλος του προηγούμενου έτους, που είναι ο νέος ειδικό εκπρόσωπος για το κέρας της Αφρικής. Τον είχαμε δεχτεί όταν ξεκίνησε. Θα αναφερθούμε στη διάσκεψη του Λονδίνου για τη Σομαλία που έγινε στο τέλος του μηνός Φεβρουαρίου. Μια πολύ σημαντική διάσκεψη, γιατί το σύνολο αυτών που εμπλέκονται στην υπόθεση της Σομαλίας ήσαν παρόντες. Αν και κάποιοι παρατηρητές πιστεύουν ότι ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης από ό,τι φαίνεται ελαχιστοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της διάσκεψης αυτής. Ο κ. Ρόντος ή το παρόν ανελήφθησαν και συγκεκριμένες υποχρεώσεις από πλευράς της κυρίας Άστον εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν εν πάση περιπτώσει γίνει προσπάθειες έτσι ώστε η αστάθεια η οποία σοβεί στη Σομαλία και η οποία θα έλεγα γεννά το φαινόμενο της πειρατείας να εκριζωθεί και μια πολιτική λύση να διαγραφεί ανάμεσα στις ε, ε, διάφορες ε, φατρίες, τις σομαλικές, είτε φατρίες περιφερικές, είτε φατρίες φιλετικές. Ξέρετε επίσης ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ξεκινήσει την EMTM, μια αποστολή στο έδαφος της Σομαλίας, μάλλον στο έδαφος της Ουγκάντα για την εκπαίδευση στρατιωτών και προσωπικού ασφαλείας της Σομαλίας. Είχε ξεκινήσει πέρυσι με ενθαρρυντικά πρώτα αποτελέσματα και με μια έκθεση η οποία μας επέτρεψε να εξελίξουμε και να βελτιώσουμε την συγκεκριμένη αποστολή. Είδαμε με ευχαρίστηση τότε ότι οι παρατηρήσεις τις οποίες είχαμε συλλέξει σαν αντιπροσωπείες συνέπιπτον με τους πολιτικούς προσανατολισμούς των ΚΟΠΣ έτσι ώστε να βελτιωθεί ακόμα περισσότερο η αποτελεσματικότητα της. Το κέρας της Αφρικής λοιπόν είναι το κατεξοχήν θα έλεγα θέατρο όπου εξελίσσεται η εξωτερική μας πολιτική και στον τομέα της ασφαλείας. Θα ξεκινήσω με τον Ναύαρχο Πότς, αν θέλετε, για το θέμα της Αταλόντ, τη UNAV4 εναντίον της πειρατείας. Πού βρισκόμαστε, Ναύαρχε, τι εξελίξεις έχουμε, πώς έχουν εξελιχθεί τα πράγματα και πώς βλέπετε την εξέλιξη της Αταλάντα στο μέλλον. Uh, uh, Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, είναι ιδιαίτερη χαρά για μένα να παρίσταμαι εδώ και να μπορέσω να συζητήσω μαζί σας και ευχαριστώ πολύ για αυτή την ευκαιρία να σας ενημερώσω για τα όσα συμβαίνουν με τη δράση Αταλάντη και τα όσα σχεδιάζουμε για το μέλλον θα σας επικαιροποιήσω, θα σας ενημερώσω με κάποιες από τις σκέψεις μας. Τι σημαίνει αυτό για τις δράσεις αυτές ε, σε σχέση με το 2012. Στρεφόμενοι στο 2011 και αυτά που έγιναν, το χαρακτηρίζω ως έτος δύο πλευρών. Κατά το πρώτο ημισή 28 σκάφη ε, ήταν θύματα πειρατείας ε, στον Ινδικό ωκεανό και στη Σομαλία. Κατά το δεύτερο ημισή του έτους μειώθηκε σε τρία μόνο αυτός ο αριθμός. Αν λοιπόν βρισκόμαστε το Μάτιο σε αυτή την αίθουσα πριν από ένα χρόνο, χρόνο θα μιλούσαμε για 33 σκάφη θύματα πειρατείας ε, προς τις ε, ακτές ε, της Σομαλίας με 750 ομήρους. Σήμερα είναι 8 αυτά τα σκάφη και 213 οι όμηροι. Πιστεύω λοιπόν ότι αυτό έχει οδηγήσει σε αλλαγές και υπάρχουν αρκετοί συντελεστές για αυτές τις αλλαγές. Πρώτον, έχουμε την αυξημένη υιοθέτηση των βέλτιστων πρακτικών διαχείρισης από πλευρά των ναυτιλιακών κύκλων. Πέρσι είδαμε ότι πήραν μέτρα αυτοπροστασίας αυτά τα σκάφη και φτάσαμε σε ένα επίπεδο πλέον <coughs> που δεν θα ε, παρεκκλίνουμε από αυτό. Και έχουμε κάποιους τομείς της αγοράς που ε, παραμένει σε σχέση με αυτά τα μέτρα αυτοπροστασίας ε, εκτός ίσως. Και βλέπουμε και αύξηση όσον αφορά την ιδιωτική ασφάλεια από τους ε, ναυτιλιακούς κύκλους. Μέχρι σήμερα 100% με επιτυχία στέφθηκαν αυτά τα μέτρα στην αποτροπή επιθέσεων. Έχουν και το όφελος για μας που δίνουν άμεσα την δυνατότητα να εντοπίσουμε και να παρακολύσουμε και να βλάψουμε τις πειρατικές δράσεις. Κατά τα τρία έτη αυτής της δράσης μάθαμε πολλά πράγματα. Πώς μπορούμε με τον καλύτερο τρόπο να αντιμετωπίσουμε πειρατές και να σταματήσουμε τη δράση τους στις ανοιχτές θάλασσες. Καθώς και πέρσι στην Ευρωπαϊκή Ένωση είχαμε πιο αποτελεσματικούς κανόνες εμπλοκής. Και για παράδειγμα τον Ιανουάριο εφέτος παράλληλα με τις ε, δυνάμεις ε, του ΝΑΤΟ και τον στρατιωτικό συνασπισμό καταφέραμε οκτώ τέτοιες ε, δράσεις με σκαφίδια από πλευράς των πειρατών να τις παρακολουθήσουμε, να τις αναχαιτήσουμε και ο τελικός συντελεστής που θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας σε αυτόν και είναι πιο δύσκολο να καταπολεμηθεί ο στοιχείο είναι η διαχείριση στην ίδια την ε, Σομαλία και η δυναμική στην Σομαλία, στην ξηρά. Όταν βλέπουμε την ε, Πούντλαντ και την Σομάλιλαντ ότι πρέπει να αναλαμβάνεται δράση κατά της πειρατείας και εκεί και είδαμε και κάποιους φυλάρχου ε, και τη δυναμική που εξελίσσεται εκεί που δημιουργεί μερικά μεγαλύτερες δυσκολίες πλέον για τους πειρατές να δρουν από εκεί. Πού βρισκόμαστε όσον αφορά την πειρατεία τώρα. Μετά από ένα έτος ρεκόρ με ε, απαιτήσει για λίτρα θα χαρακτήριζα τους ε, ε, πειρατές ότι έχουν αποκομίσει ωφέλη και βρίσκονται τώρα σε αυτή την κατάσταση που επωφελήθηκαν και τώρα με την περίοδο των ε, μουσώνων που ε, πρόκειται να ξεκινήσει και αυτή η περίοδος θα ξεκινήσει μέχρι τον Ιούνιο όπου ε, έχουμε, θα έχουμε τους νοτιοδυτικούς μουσώνες και είναι πολύ δύσκολο να δρουν υπό αυτές τις προϋποθέσεις. Θα προσπαθήσουν να ανακάμψουν και να αυξήσουν το δυναμικό τους αν, μια και πρόκειται για μια εγκληματική επιχείρηση που θα βρεθεί με, υπομεγάλη πίεση τελικά. Ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας στην, στο στρατηγικό πλαίσιο έχουμε τακτικής φύσεως επιτυχίες μέχρι σήμερα. Όμως το δυναμικό των πειρατών εξακολουθεί να υφίσταται επειδή δεν υπάρχει σωστή διακυβέρνηση στην ξηρά και ο τρόπος ε, δράσης των πειρατών δείχνει ότι μπορούν να προσαρμόζονται γρήγορα, αλλάζει ο τρόπος δράσης τους ε, και μπορούν ε, να δράσουν και αυτό είναι συνέχεια απειλή. Δύο συμπεράσματα μπορώ να συναγάγω από αυτές τις δράσεις μας. Πρώτον, τώρα είναι η χρονική στιγμή να αυξήσουμε την πίεση και δεύτερον, τώρα είναι η χρονική στιγμή να συνεργαστούμε με τους ίδιους τους Σομαλούς επικοδομητικά. Και εδώ βρίσκεται ο ρόλος κλειδιού που έχει ο ύπατος ε, εκπρόσωπος, ύπατος απεσταλμένος. Και έχει τεράστια σημασία αυτή η αποστολή του για το συντονισμό με τους Σομαλούς. Πώς θα αυξήσουμε την πίεση στους πειρατές πρώτο το πρότυπο επιχείρησης ή δράσης, αυτό είναι που χρησιμοποιούμε γιατί είναι εγκληματική οικονομική δραστηριότητα αυτή και είναι σχετικά απλό να την κατανοήσει κανείς. Ξεκινάμε τη συλλογή κονδυλίων, μετά υπάρχουν οι επενδύσεις, οι πειρατές μετά προετοιμάζουν στην ξηρά και στην, ε, στην παράκτια περιοχή ε, τα όπλα τους και τις δυνατότητές τους, ε, βγαίνουν στην, στον, στη θάλασσα, επιστρέφουν και μετά έχουμε την διασπορά των κονδυλίων που έχουν συλλεγεί και επανεπενδύονται σε επιχειρηματικές δράσεις. Αυτή τη στιγμή σε σχέση με στρατιωτική πτυχή η δράση μας επικεντρώνεται κυρίως στη φάση στη θάλασσα, στην ανοιχτή θάλασσα. Βλέπουμε πώς μπορούμε να δράσουμε και κατά των άλλων συνιστοσών αυτού του προτύπου επιχείρησης των πειρατών και κατά την μέσα μεσολαβητική περίοδο μεταξύ των μουσώνων θα πρέπει να αυξηθεί η πίεση στις παράκτιες περιοχές εκεί όπου ε, υπάρχει η μεγαλύτερη επιτυχία για αυτούς αλλά και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε επιπρόσθετα ώστε να δυσχεράνουμε ακόμα περισσότερο για αυτούς να μπορούν να ε, φεύγουν από τις έδρες τους και να κάνουν αυτές τις επιθέσεις. Τους τελευταίους μήνες εξετάσαμε εκ του σύνεγγυς με τις αρχές της Σομαλίας και έχουμε εμπλακεί όχι μόνο με την προσωρινή ομοσπονδιακή κυβέρνηση αλλά και σε υπουργικό επίπεδο και επίσημο επίπεδο με την ίδια την Πούντλαντ, τους ε, κυβερνητικούς αξιωματούχους ε, και είμαστε με στεναρό πείσμα αποφασισμένοι οποιαδήποτε δράση θα αναλυθεί να μην διακυβεύει άλλες δράσεις όσον όσον αφορά την ασφάλεια, την ανάπτυξη, την ανθρωπιστική βοήθεια που παρέχεται προς τη Σομαλία. Επίσης προσέχουμε ιδιαίτερα να λάβουμε ιδιαίτερα σοβαρά τις απειλές όσον αφορά τους ομήρους και θα πρέπει πραγματικά να μην αυξάνονται οι κίνδυνοι έναντι των ομήρων, να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Με οποιαδήποτε δράση, στα πρώτα δυόμιση χρόνια αυτών των δράσεων, είμαστε, αντιδρούσαμε απλά σαν όσα έκαναν οι πειρατές. Θέλουμε όμως τώρα να είμαστε ενεργητικοί οι ίδιοι και όχι μόνο να αντιδρούμε στις δράσεις των πειρατών. Αυτό εξαρτάται βέβαια από την συνειδητοποίηση, το κατά πόσο θα έχουμε συνειδητοποιήσει πλήρως ε, όλες τις συνιστώσεις και το επίπεδο ελέγχου χωρίς να υπησέθω σε λεπτομέρειες λειτουργικές των δράσεών μας. Είμαστε στεναρά αποφασισμένοι η διαδικασία λήψεως αποφάσεων να εξετάζεται με τον σωστό τρόπο και σε βάθος ώστε να διασφαλίζουμε ότι οι ύψιστες αυτές στρατηγικές προτεραιότητες θα λαμβάνονται υπόψη από πλευρά μας. Στρεφόμενοι προς το μέλλον. Είμαι πεισμένος ότι ο ρόλος μας είναι πραγματικά να αντιμετωπίσουμε τα συμπτώματα μιας αποτυχημένης ε, στη διακυβέρνησή της χώρας. Για να αντιμετωπίσουμε στα αίτια, στη ρίζα του το κακό πρέπει να αυξήσουμε τη σωστή διακυβέρνηση και την ασφάλεια όσον αφορά αυτή τη χώρα. Αναγνωρίζω βέβαια ότι ο ρόλος αυτός είναι ρόλος άλλων πέρα από τον δικό μου ρόλο και τον δικό που είμαστε στρατιωτικοί και ασχολούμεθα με την ε, στρατιωτική δράση σε αυτό το επίπεδο. Σαν συνέπεια υποστηρίζουμε στενά τις δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδιαίτερα τον ειδικό απεσταλμένο και την αποστολή του, αλλά στρεφόμαστε και προς την μελλοντική δράση για το Regional Capacity Building, την αύξηση του περιφερειακού δυναμικού και την υποστήριξη αυτού του δυναμικού και την παροχή υποστήριξη στους Σομαλούς και στο Γκάρμαντου και το Πούντλαντ που είναι περιοχές από τις οποίες δρούν κυρίως οι πειρατές. Υπό τους όρους της τέταρτης γενεάς έχουμε και μία διάσκεψη κατά τις αρχές αυτού του μήνα και μπορώ να αναφέρω ότι σε σχέση με το 2012 και την προέκταση αυτών των δράσεων μέχρι το 2013, παρόλη την διάρκεια επί τρία έτη αυτής της δράσης και υπάρχει βέβαια μεγάλη πίεση όσον αφορά τα δημοσιονομικά και τα κονδύλια από τα κράτη-μέλη, πρέπει να διασφαλιστεί η λειτουργικότητά μας. Υπάρχουν στοιχεία κλειδιά που θέλουμε να αυξηθεί η χρηματοδότηση για να είμαστε λειτουργικοί και δεν είμαστε καθόλου αυτοικανοποιημένοι και δεν εφησυχάζουμε καθόλου όσον αφορά τα όσα έχουν γίνει. Σε σχέση όμως με το που βρισκόμαστε, σε σχέση με τον προηγούμενο χειμώνα, όπου ήταν πολύ χαμηλές οι ισροές, στρεφόμαστε προς το μέλλον με ελπίδες ότι θα βελτιωθούν τα πράγματα εφέτος και εφεξής Και κάποια σχόλια όσον αφορά το μέρος εκείνο της αποστολής μας που ήταν ε, εκείνο το οποίο λειτουργήσε ως καταλήτης ε, για να είμαστε αποτελεσματικοί και η υποστήριξη του ε, Παγκόσμιου Επισητιστικού Προγράμματος ε, και της Διασφάλισης Ανθρωπιστικής Βοήθειας. Το 2011 το Παγκόσμιο Επισητιστικό Πρόγραμμα 35.000 τόνοι μεταφέρθηκαν από πλευρά τροφίμων σε αυτή την περιοχή. Μέχρι το Δεκέμβριο είχε αυξηθεί σε πάνω από 90.000 τόνους ε, αυτή η ποσότητα. Αυτό το πρόγραμμα που πρέπει να διασφαλιστεί πρέπει να μπορέσει να συνεχιστεί. Το τι συνέβη κατά τους τελευταίους 4-5 μήνες πρέπει να εξεταστεί σε στενή διασύνδεση με τα όσα κάνουμε εμείς και με το, τα όσα κάνει το ε, Παγκόσμιο Επισητιστικό Πρόγραμμα. Η φιλοσοφική μας προσέγγιση άλλαξε από την παροχή... Ε, ασφάλεια στις νιοπομπές θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι θα είναι επαρκώς προστατευόμενα αυτά τα πλοία και θα προστατεύονται επαρκώς όπου και να βρίσκονται και να δρούν. Και σε σχέση με αυτό το οποίο αποκαλούμε Autonomous Vessel Protection Detachments, ομάδες, αυτόνομες ομάδες προστασίας σκαφών και που πρέπει έτσι να μπορούν να βοηθούν και την ροή εμπορευμάτων και ε, αγαθών στο επισητιστικό πρόγραμμα βοήθειας. Το τι συνέβη σε σχέση με την απουσία ε, δυναμικού έχει οδηγήσει στον πολλαπλασιασμό των συντελεστών αυτών. Πρέπει να είμαστε αποτελεσματικοί στην αποτροπή και αναχέτηση των δράσεων των πειρατών. Έχουμε τώρα μια Ολλανδική τέτοια αυτόνομη ομάδα προστασίας που δρά σε ένα, όσον αφορά και πλοίο το οποίο έχει χρονοναυλωθεί για αυτή την επισητιστική βοήθεια και πρέπει να δούμε ότι πολλαπλασιάζονται αυτές οι πρωτοβουλίες Σαν συνέπεια όλων αυτών, από τακτικής πλευράς έχουμε σημειώσει πρόοδο. Σίγουρα η δυναμική αύξηση που είδαμε να σημειώνεται από το 2008 έχει μετριαστεί τώρα πλέον η αυξητική αυτή τάση και με τους ναυτιλιακούς κύκλους και τις δράσεις που αναλαμβάνουν προσπαθούμε να αναχαιτήσουμε τις ε, ε, πειρατείες. Και όταν λέω εμείς, ε, εμείς και όσον αφορά τις δικές μας δράσεις και τους άλλους που εμπλέκονται με τις δράσεις αυτές. Πρέπει να αντιμετωπιστούν όμως τα αίτια του κακού, στη ρίζα τους και αυτά βρίσκονται στην ανασφάλεια και στην κακή διακυβέρνηση όσον αφορά την ίδια την στεριά, δηλαδή στη Σομαλία. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή την παρουσίαση. Πιστεύω ότι ορισμένοι συνάδελφοι θα θέσουν κάποια ερωτήματα σε σχέση με τα διάφορα σημεία τα οποία θέσατε. Θα ήθελα να επανέλθουμε σε ένα πρόβλημα το οποίο αναφέρατε, αλλά θα ήθελα να πούμε περισσότερες λεπτομέρειες ή δυνατόν όσον αφορά το δυναμικό, τις δυνατότητες. Γιατί πρόκειται για μία από τους βασικούς λόγους ενσχύσεων αφορά την καλή λειτουργία ε, δηλαδή να υπάρχουν επαρκή μέσα ε, ναυτικά ή ε, εξαίρως όσον αφορά τη συμμετοχή των διαφόρων ευρωπαϊκών ε, δυνάμεων και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν να κινητοποιήσουν τις δυνάμεις της εάν μπορείτε δηλαδή να μας κάνετε κάποιες διευκρινήσεις σε σχέση με αυτά τα σημεία. Είναι κάτι το οποίο σας ε, ανησυχεί ή μπορείτε να αντιμετωπίσετε τις ε, προκλήσεις ε, της, που θα έχουμε την άνοιξη. Ο κύριος Γκάλερ θέλει να πάρει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Νάβαρχε. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσίασή σας. Ο κύριος ε, Πρόεδρος ανέφερε, προανέφερε μία από τις ερωτήσεις που εγώ ίδιος θα έθετα όσον αφορά την, ε, την έκταση των μέσων που χρειαζόμαστε και αυτά τα μέσα που έχουμε πραγματικά στη διάθεσή μας εκεί. Ε, νομίζω ότι είναι σημαντικό να μας το εξηγήσετε, ίσως στο συνολικό πλαίσιο έχουμε τη συμμετοχή του ΝΑΤΟ και ίσως ε, θα μπορούσατε να μας πείτε κάποια πράγματα εν σχέση με το πώς αναπτύσσεται η συνεργασία με τρίτες χώρες, την Κίνα, την Ινδία ή τη Ρωσία. Γιατί εδώ ε, ακούμε ότι υπάρχουν ε, κάποιες αποστολές, αποστολές που συνεργάζονται με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, νομίζω ότι από πολιτική άποψη θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο πρώτος στόχος έχει επιτευχθεί, δηλαδή ε, θέλουμε ε, μέσω του Παγκόσμιου Επιστημιστικού Προγράμματος να εξασφαλίσουμε ούτω ώστε όλες οι αποστολές στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος να φτάνουν στο στόχο τους. Και νομίζω ότι αυτή, αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό μήνυμα το οποίο μπορούμε να διαδώσουμε διεθνώς. Ε, θεωρώ ότι τα συμπεράσματα στα οποία καταλήξατε, δηλαδή ότι ήρθε το πλήρωμα του χρόνου να αυξήσουμε την πίεση, ε, μπορεί να πετύχει μόνο εάν έχουμε αυξήσει τις ε, δυνατότητές μας, το δυναμικό μας. Την ε, Πέμπτη είναι το Συμβούλιο των Υπουργών Άμυνας και αυτή θα ήταν και ερώτησή μας. Τι θα μπορούσατε να διατυπώσετε ως αίτημα προς τους πολιτικούς γιατί εμείς, ε, για να μπορούμε να σε επιστηρίξουμε και εμείς από τη δική μας την κοινοβουλευτική πλευρά. Τώρα, τα ερωτήματα τα οποία τίθενται βεβαίως ε, σχετίζονται με, το, με την εμβέλεια αυτών των χερσαίων επιχειρήσεων, για παράδειγμα. Πώς θα μπορούσε κανείς να τις ε, διευρύνει στην ξηρά. δηλαδή, ούτως ώστε να μπορούν να φτάσουν οι πειρατές εύκολα στην ξηρά. Ε, αυτή όμω είναι και μια πολιτική απόφαση. Πώς θα μπορούσε να τροποποιηθεί, να διευρυνθεί ενδεχομένω σχετική εντολή. Η δική μου τεχνική ερώτηση είναι η εξή. Έχουμε τη δυνατότητα από μεγάλη απόσταση να, μπορούμε, να μπορέσουμε να επιτεθούμε σε αυτές τις... Ε, όταν φτάνουν στην ξηρά ή ε, θα πρέπει να κινηθούμε πράγματι μόνο εξαέρος με τα ελικόπτερα ε, αντιμετωπίζει το κίνδυνο τελικά να μπορέσουν να περάσουν από την, να φτάσουν στην ξηρά. Ε, αυτά είναι θέματα που αφορούν τη διεύρυνση της επιχειρησιακής εντολής. Ευχαριστούμε πολύ ο κύριος Σίμκε. panu, panie admirale, za bardzo ciekawą informację. Mm, z danych, które pan przekazał, wynika, że sytuacja na szczęście się poprawia. Έχω την αίσθηση ότι η κατάσταση έχει αρχίσει να βελτιώνεται. Η βελτίωση της κατάστασης οφείλεται σε τρεις παράγοντες και όχι μόνο στη στρατιωτική, ε, καθαρά στρατιωτική δραστηριότητα. Το πρώτο είναι η μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα του συνόλου των δραστηριοτήτων μας στην περιοχή. Αναφερθήκατε σε αυτό. Αναφερθήκατε επίσης και στον διαφορετικό τρόπο που αντιμετωπίζει το θέμα ο εφοπλιστικός κόσμος. Ε, προσπαθούν τα πλοία του συγκεκριμένου του χώρου να προστατεύονται ε, και τα ίδια. Δεύτερον, έχουν εξελιχθεί κάπως τα πράγματα στη Σομαλία και αυτό οδηγεί στη βελτίωση της κατάστασης. Αυτό το οποίο πραγματικά με ανησυχεί σε αυτή τη φάση είναι το θέμα το οποίο έθεσε ξεκάθαρα ο κύριος Ντονζόν. Είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να μας απασχολήσει. Είσαστε ο υπεύθυνος μιας στρατιωτικής αποστολής και έχετε στη διάθεσή σας συγκεκριμένες ναυτικές μάχημες μονάδες. Συζητήσαμε το θέμα αυτό στο Στρασβούργο την προηγούμενη εβδομάδα, προετοιμαστήκαμε ελπίζω σωστά και δεν ξέρω αν κατανόησα καλά τα εξή στοιχεία. Λέγουν τα στοιχεία, το 2009 υπήρχαν 35 σκάφη. Πέρυσι ήταν 10 τα σκάφη και φέτος έχετε στη διάθεσή σας μόνο τρία σκάφη. Εάν αλήθεια είναι αυτό που είπα, τότε το μήνυμα είναι πολύ κακό. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς έχει μειωθεί δια 10 ε, ο αριθμός ο οποίος ξεκίνησε, ο αριθμός των πλοίων με τα οποία ξεκινήσατε. Και έτσι και αλλιώ ο αριθμός των τριών σκαφών είναι κάτι το οποίο θα έλεγα σε επίπεδο στρατιωτικών ικανοτήτων είναι ιδιαίτερα αποδυναμωμένο. Λοιπόν, το επόμενο ερώτημα πρόκειται για την Αταλάντα. Όπως είπα είναι μια επιχείρηση η οποία διεξάγεται στα πλαίσια της εξωτερικής δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διασφάλιση της ειρήνης και της ασφάλειας στην περιοχή. Και θα ήθελα να θέσω το ερώτημα στον Άβαρχο Πότς. Ε, στην καταπολέμηση της πειρατείας ε, έχουν πραγματικά εμπλακεί οι Ρώσοι και οι Κινέζοι. Οι Ρώσοι ε, κάτι τέτοιο έλεγαν. Υπάρχει λοιπόν στρατιωτική δύναμη ρωσική και κινέζικη στην περιοχή σας και αν ναι έχετε τη δυνατότητα συνεργασίας με αυτούς, κυρία Νικολαή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχω δύο ερωτήσεις. Η πρώτη σχετίζεται με την ε, συνεργασία σας με τα με δυνατότητες ιδιωτικής ασφάλειας, με ιδιωτικά σκάφη γιατί υπάρχουν πολλοί από εσά που χρησιμοποιούν ιδιωτικέ εταιρείε, υπάρχει ένα τέτοιο είδο συνεργασία και πώ αντιμετωπίζετε αυτή τη μορφή συνεργασία από τη δική σα πλευρά. Η δεύτερη ερώτηση συνδέεται με την εντολή σα, γιατί όταν ήμουν στο Τζιμπουτί, πολλοί ε, αξιωματούχοι μας είπαν ότι δεν είναι ευτυχεί για τις ε, δυνατότητες που τους παρέχει η εντολή τους τώρα έχετε, τη δυνατότητα να, έχετε τώρα τη δυνατότητα να παρεμβαίνετε σε όλες τις καταστάσεις. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Κρόνμπεργκ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για το γεγονός ότι η πειρατεία μπόρεσε να αναχαιτιστεί, όπως αναφέρατε. Αναφέρεται επίση το θέμα των βασικών αιτίων καθώ και τη διακυβέρνηση και τη ασφάλεια. Μπορείτε να δείτε κάποιες, ε, βλέπετε κάποιε αλλαγέ όσον αφορά αυτά τα θέματα κατά τη διάρκεια δική δικής θητείας. Όσον αφορά δε τη διεύρυνση τη ε, Ατλάντα, Αταλάντα, ε, πώς αντιμετωπίζετε του κίνδυνου που συνδέονται με αυτήν. Για παράδειγμα, εάν οι πειρατέ εγκατασταθούν σε επικοινωνικατοικημένε περιοχέ, για παράδειγμα. Τέλος, ε, βλέπ, όσον αφορά τον αριθμό των πειρατών, δηλαδή των νέων ανθρώπων που αυξάνεται, γιατί διάβασα μια σχετική μελέτη όταν ε, ρωτήθηκαν τι θέλουν να κάνουν οι νέοι άνδρες στη Σομαλία, απαντούσαν ότι θέλουν να γίνουν πειρατές. Εάν αυτό λοιπόν, ε, αυτή είναι η μελλοντική απασχόληση των νέων στη Σομαλία, πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση, ούτως ώστε να μειωθεί αυτό το κίνητρο. Ο κύριος Στάνακα, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να χαιρετήσω εκπροσωπώ μια περιοχή όπου έχει την έδρα στον Όρφογκ. Επίσης είμαι εισηγητής του Κοινοβουλίου για το κέρας της Αφρικής. Θα ήθελα λοιπόν να δώσετε κάποιε συμβουλές για τη δική σας έκθεση. Θα θέσω λοιπόν μια σειρά ερωτήσεων. Ε, η πρώτη καλύφθηκε. Σε ποιο βαθμό θέλετε να διευρυνθεί η εντολή, το εύρο εντολή σας για τις επιχειρήσεις σα. Εγώ θα ήθελα να υπάρξει το δικαίωμα να πάει κανείς ε, στην, ε, στην ξηρά, ώστε να μειωθούν οι δυνατότητες των πειρατών. Ε, νομίζω ότι θα ήταν εξαιρετικά χρήσιμη αυτή η διεύρυνση της εντολής. Ίσως μια συμφωνία συνεργασίας με την ΑΜΙΣΟΜ να μπορούσε να γίνει σε αυτήν την κατεύθυνση. Η δεύτερη ερώτηση επίσης ε, τέθηκε όσον αφορά των εμπορικών ε, ιδιωτικών σκαφών που καλύπτουν θέματα ασφαλείας. Μέχρι στιγμής εγώ ξέρω μόνο ένα παράδειγμα ενός σκάφου το οποίο εχμαλωτίστηκε και ορισμένες, όπου υπήρχε κάποιο προσωπικό Ε, ορισμένες ε, χώρες ε, το επιτρέπουν, άλλες ε, όχι. Αυτή τη συμμετοχή του δικού του εμπορικού στόλου σε τέτοιου είδου επιχειρήσει. Χθε είχα μια συνάντηση, γιατί είμαι hands they Στην Επιτροπή με την ε, Ταϊβάν ε, υπάρχει δυνατότητα συνεργασίας με την ε, Κίνα ούτως ώστε να συμμετάσχουν κάποια κινέζικα σκάφη σε τέτοιου είδους επιχειρήσεις. Ε, υπάρχουν, ίσως υπάρχουν τέτοιου είδους δυνατότητες συνεργασίας γιατί τα δικά τους ε, αλευτικά σκάφη πολύ συχνά γίνονται στόχος ε, επιθέσεων. Οχτώ πλοία του κινέζικου στόλου έπεσαν ε, θύματα, αλευτικά σκάφη. Και συμφωνείτε τελικά η επιχείρηση Αταλάντα να συνεργαστεί με ειδικά σκάφη ή με άλλα σκάφη τρίτων χωρών. Μιλούσα να υπάρξει μια σπίδα προστασίας Τέλος και πάλι θα ήθελα να πω ότι είμαι υποστηρικτής της αναγνώρισης του Σομάλι Λαντ που ήταν μια παλιά βρετανική απικία και έγινε μια συνδιάσκεψη στο Λονδίνο για τη Σομαλία. Το Σομάλι Λαντ υπήρξε εξαιρετικά βοηθητικό όσον αφορά την καταπολέμηση τη υπηρετία και χρειάζεται περισσότερη ενίσχυση τη δική του ακτοφυλακή. Υπάρχουν κάποιε επαφέ και διερεύνηση αυτού του θέματο. Εγώ ε, όσον αφορά τις ε, φυλακές, ε, στη Βρετανία υπάρχει μια απαγόρευση δημιουργίας φυλακών στην περιοχή αυτή. Ποιος πρόκειται, θα πρέπει οι πειρατές να φυλακίζονται, αλλά πώς θα εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση. Γιατί υπάρχουν κάποια προβλήματα σε σχέση με τις περικοπές του προϋπολογισμού και την νομιμότητα της δημιουργίας φυλακών από κοινοτικά κονδύλια. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας καλωσορίζω, λοιπόν, κύριε Πότς, και σας ευχαριστώ για την ομιλία σας. Σας συγχαίρω γιατί έχει βελτιωθεί κατά πολύ η κατάσταση, παρότι υπάρχει το πρόβλημα. Αναφερθήκατε ότι εσείς συγκεντρώνετε την προσοχή σας στις θαλάσσιες επιχειρήσεις. Είπατε όμως ότι φέτος ίσως να στοχεύσετε λίγο και στις παράκτιες περιοχές. Και θα μπορούσατε λοιπόν να μας δώσετε κάποιες περισσότερες λεπτομέρειες γύρω από αυτό. Ξέρουμε ότι το βασικό πρόβλημα είναι η κρατική δυσλειτουργία της Σομαλίας. Ο ε, κρατικός μηχανισμός στην ουσία είναι στο μηδέν. Ε, πότε πιστεύετε ότι θα υπάρξει μια ανόρθωση της κατάστασης εκεί. Ευχαριστώ κυρία Σαρζεντίνη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχω δύο ερωτήσεις. Καταρχάς, σε σχέση με αυτά τα οποία έλεγε μόλις ο κύριος Γκάλερ για την στρατιωτική παρουσία πλέον α, στο, όχι μόνο στη θάλασσα αλλά και στις παράκτιες περιοχές. Θα ήθελα λοιπόν να μας δώσετε λίγα περισσότερα στοιχεία ε, γι' αυτό. Έχουμε κάποιες αμφιβολίες σχετικά με τα πιθανά αποτελέσματα αυτής της εμπλοκής. Έχουμε φόβους να δούμε τα πράγματα να κλιμακώνονται σε επίπεδο βίας. Και θα ήθελα να αναφερθείτε λίγο και στα θέματα της παράνομης αλίας. Αν κατάλαβα καλά, ένας από τους στόχους τους οποίους έχετε είναι και η καταπολέμηση της παράνομης αλλιευτικής δραστηριότητας. Τι αποτελέσματα είχατε ως προς αυτό. Ευχαριστώ. Ο Ναύαρχος έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ για όλες αυτές τις ερωτήσεις σας και θα προσπαθήσω να τις συστηματοποιήσω μία προς μία στις απαντήσεις μου. Υπάρχουν αρκετές ερωτήσεις αν έχουμε επαρκείς πόρους για αυτή την αποστολή μας. Πρώτα απ' όλα, μέσα σε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο, ο δικός μου τομέας δράσης και από την, τον, τον Ατλαντικό ως τα Ουράλια και από την Μεσόγειο μέχρι αυτή την περιοχή. Έχουμε τεράστιο πεδίο δραστηριοτήτων και ως στρατιωτικός ηγέτης, ως επικεφαλής θα θέλαμε να έχουμε τις μέγιστες στρατιωτικές δυνάμεις. Ακόμα και αν έχουμε ε, αυτές τις ε, δυνάμεις στη διάθεσή μας, πάντα υπάρχει επαρκές πεδίο για τη δράση τους. Έχει αρκετά δημοσιοποιηθεί ότι κατά τη διάρκεια αυτού του χειμώνα είχαμε χωρίς προηγούμενο πολύ ε, χαμηλό επίπεδο και αυτό οδηγεί σε μια ανάκαμψη τώρα. Αν δει κανείς το 2012 για τον αριθμό αυτό των δυνάμεών μας είναι καλύτερο το αποτέλεσμα από ό,τι συνέβαινε το 2011. Επανερχόμαστε στα επίπεδα που είχαμε όταν ξεκίνησε αυτή η δράση. Ένα άλλο σημείο που θα ήθελα να αναφέρω, δεν συμβαίνει πάντα κατά τη διάρκεια του έτους. Έχουμε και τις, ε, τους βορειοανατολικούς και νοτιοδυτικούς μουσώνες. Ε, κατά τους ε, νοτιοδυτικούς από τον Ιούνιο στα τέλη Σεπτεμβρίου υπάρχει αυτή η επίπτωση. Και όσον αφορά τα μικρά σκάφη που βγαίνουν στην ανοιχτή θάλασσα δυσκολεύονται πολύ οι προϋποθέσεις για αυτά. Η περίοδη εχμής για την πειρατεία που από τον Οκτώβριο στο Δεκέμβριο και στην περίοδο του Ιουνίου είναι εκείνες που πρέπει να συνεργαζόμαστε με τα κράτη που συνεισφέρουν ώστε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Πάντα μπορούμε να έχουμε περισσότερες δυνάμεις αλλά σε ρεαλιστικό πλαίσιο με τις δυνάμεις που μας διατίθενται έχουμε το ελάχιστο αναγκαίο για να ανταποκριθούμε στις υποχρεώσεις μας πιστεύω και επιπλέον γι' αυτό κάποιες ερωτήσεις ε, για το πώς συνεργαζόμαστε και με το ΝΑΤΟ και ανεξάρτητους ε, εμπλεκόμενους. Θα έλεγα ως στρατιωτικός ε, και όταν πέρσι ξεκίνησε αυτή η δράση και την ανέλαβα βλέποντας το σύνθετο και περίπλοκο της δομής ε, από πλευράς στρατιωτικών δράσεων με τρεις διαφορετικούς οργανισμούς που είχαν αναλάβει αυτές τις δράσεις είπαμε ότι θα ήταν ένα δύσκολο πλαίσιο να λειτουργήσουμε έτσι. Στην πρακτική εφαρμογή όμως είναι πολύ πιο απλά τα πράγματα από ό,τι φαίνονται σε με αυτή την προσέγγιση. Το επίπεδο στην τακτική συνεργασία είναι χωρίς προηγούμενο θα έλεγα υποστατιωτικούς όρους σε καθημερινή βάση και στις, ε, ε, στα, στο επιτελείο μας αλλά και στο ε, ε, επιτελείο των άμεσων δράσεων επιτόπου υπάρχει μια χωρίς καμία καμπή ή ρήξη ροή πληροφοριών και για την, ε, ε, τα όσα συμβαίνουν στην Σομαλία και σε καθημερινή βάση συντονίζουμε τις δραστηριότητες μας. Παρόμοια όταν συμβαίνουν κάποια συμβάντα και πρέπει να αντιμετωπίσουμε και να αντιδράσουμε άμεσα έχουμε ένα σύστημα κοινό σύστημα επικοινωνίας που επιτρέπει όχι μόνο σε εμά στο ΝΑΤΟ και στις συνασπισμένες ε, θαλάσσιες δυνάμεις να ανταλλάσσουν πληροφορίες αλλά και με την πρωτοβουλία Mercury, Ερμής υπό την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε και τους ανεξάρτητους που εντάσσονται σε αυτό το πλαίσιο και τους Ρώσους και τους Κινέζους, τους Ιάπωνες αλλά επίσης και περιφερειακές χώρες που συνεργάζονται και εντάσσονται εκεί. Γενικά πιστεύω ότι το επίπεδο συνεργασίας και συντονισμού βρίσκεται σε πολύ ψηλό επίπεδο και έτσι α, έχουμε ένα πολύ καλό επίπεδο τακτικής συνέργειας στις λειτουργικές μας δράσεις στην περιοχή αυτή. Κάνοντας λόγο για την συνεργασία υπάρχουν συγκεκριμένα θέματα για την Ρωσία και την Κίνα από κοινού είναι αξιόλογο να δούμε ότι στους τρεις άξονες αυτού του συνασπισμού Ευρωπαϊκή Ένωση, ΝΑΤΟ και την Αμερικανική Συμμαχική Δύναμη αυτό το οποίο διαφοροποιεί αυτές τις συνιστώσεις από άλλες είναι ότι ουσιαστικά ουσιαστικά παρέχουμε υπηρεσίες σε όσους έχουν ανάγκη αυτές τις υπηρεσίες χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη τη σημαία τους ή την εθνικότητά τους όπως και στην ε, ναυτιλία γενικότερα. Άλλοι οι οποίοι δρούν σε αυτή την περιοχή ε, ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για τη δική τους σημαία ή της δικής τους εθνικότητας σκάφη. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν αντιδρούν και δεν συνεργάζονται όταν πρόκειται για μια κοινή δράση αλλά υπάρχει μια διαφοροποίηση όσον αφορά την προσέγγιση του και την αντιμετώπιση της πειρατείας. Και πρέπει να υπάρχει ένας ευδιάκριτος χαρακτήρας που θα ε, δρά ως στοιχείο αποτροπής για τους πειρατές και για τις δράσεις της ε, παγκόσμιας επισητιστικής βοήθειας που βρίσκεται υπό εξέλιξη και συνεχίζεται. Είναι η δράση καταλήτης σε σχέση με όλους όσους εμπλέκονται. Χρειάζεται, υπάρχει τεράστια ανάγκη να προστατεύεται αυτό το παγκόσμιο πρόγραμμα επισητιστικής βοήθειας. Έχει ανώτατη προτεραιότητα για μένα να διασφαλίσω αυτή την ασφάλεια. Αυτό το οποίο αλλάζει σε σχέση με τις απαιτήσει ε, είναι όσον αφορά τον χειμώνα η ανάγκη να προσαρμοστούμε στις, ε, στο δυναμικό που έχουμε στη διάθεσή μας και θα ήθελα να υπάρξει η δυνατότητα οι μονάδες αυτόνομης προστασίας ε, η πρώτη που ξεκίνησε τον Ιανουάριο να μπορέσουμε να δράσουμε με πολύ πιο αποτελεσματικό τρόπο παρέχοντας επαρκή, επαρκές επίπεδο προστασίας σε σχέση πάντα με το δυναμικό για παράδειγμα σε σχέση με ελικόπτερα ή ε, δράσεις που μπορεί να ε, παρέχονται από πολεμικά σκάφη ώστε να είμαστε αποτελεσματικοί και πιστικοί στην αποτροπή τη, στη δράση μας κατά της πειρατείας. Τώρα, για το αν μπορούμε να επεκταθούμε στην ξηρά ως ε, επικεφαλής στρατιωτικός κάνω για αυτά τα θέματα. Το πρότυπο προσέγγισης ξεκινά με την χρηματοδότηση, τις προμήθειες ε, και στο τέλος με την ε, αντιμετώπιση του θέματος των λύτρων. Για την πειρατεία αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να αντιδράσουμε στο σύνολο αυτών των συνιστοσών και να τις υπονομεύσουμε με δράσεις πέρα από το στρατιωτικό πεδίο και να δράσουμε όσον αφορά τη χρηματοδότηση που πρέπει να αντιμετωπιστεί Υποστηρίζω βέβαια απόλυτα ότι άλλοι πρέπει να επικεντρωθούν σε αυτό το έργο, αλλά μάλιστα θα θέλαμε να αναλυφθεί δράση σε πολύ στενή συνεργασία με τους άλλους για να καταπολεμηθούν αυτές οι, αυτοί οι συντελεστές. Πρέπει να το κάνουμε αυτό με πολύ συνετό και προσεκτικό τρόπο εστιαζόμαστε σε αυτό παρότι έχουμε στρατιωτική προτεραιότητα στη δράση μας συνειδητοποιούμε ότι έχουμε παραπληρωματικό ρόλο που επιτελούμε εδώ συμπληρωματικό ρόλο και υπάρχουν σημαντικοί περιορισμοί και όσον αφορά το επίπεδο δυνάμεων που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε όσον αφορά την επιβολή, την ε, υλοποίηση αυτών των μέτρων. Οποιαδήποτε δράση που θα αναλαμβάνουμε πρέπει να συγχρονίζεται απόλυτα με τις άλλες γραμμές δράσης ε, για την ασφάλεια, την ανάπτυξη και την ανθρωπιστική βοήθεια πολλαπλά και γι' αυτό συνεργαζόμαστε εκ του σύνεγγυς με τον ειδικό απεσταλμένο και τα άλλα όργανα και θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης ώστε να μην υπονομεύεται η δράση τους. Είναι επίσης πολύ σημαντικό να δούμε ποια είναι η εικόνα που αντανακλάται στη Σομαλία από αυτές τις δράσεις από πλευράς μας. οποιαδήποτε δράση θα αναλαμβάνουμε θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικά σταθμισμένη όσον αφορά την αναλογικότητα και το αποτέλεσμά της και πρέπει όλο και περισσότερο με τους Σομαλούς να βλέπουμε αυτές τις δράσεις. Κατά τους τελευταίους έξι μήνες συζητούμε πως ανέφερα αυτά τα θέματα μαζί τους. Υπάρχει υποστήριξη και πρέπει να υπάρχει αυτή η υποστήριξη των μέτρων αυτών. Και στην προσέγγιση αυτής της ε, περιοχής ε, διαπίστωσα σε σχέση με τους Σομαλούς όχι μόνο με την αναδυόμενη πολιτική τάξη αλλά και τους ίδιους τους Σομαλούς ότι η ανοχή τους έναντι των πειρατών μειώνεται. Ναι φυσικά ένα από τα θέματα είναι αυτοί οι νέοι που θέλουν να γίνουν μέρος και να συμμετάσχουν σε αυτές τις συμμορίες. Είναι ένα πρόβλημα αυτό διότι τους ε, θέλει και τους προσελκύει αλλά σε σχέση και με την Σομαλία, την κοινωνία της Σομαλίας βλέπουμε τις κοινότητες ε, που επιθυμούν πλέον να εκτοπίσουν αυτούς τους ε, πειρατές και να τους αποπέμψουν και πρέπει να συνεισφέρουμε στη δράση μας υπέρ αυτής της τάσης και όχι να την υπονομεύσουμε. Νομίζω, νομίζω κάλυψα τις συγκεκριμένες ερωτήσεις για τα θέματα Ρωσίας και Κίνας. Το θέμα συνεργασία τώρα με ιδιωτικές, ε, ιδιωτικούς φορείς ασφάλειας. Φυσικά τώρα για τα ε, σκάφη και την σημαία τους είναι αρμοδιότητα των κρατών αυτών ε, να δουν τι θα κάνουν είναι κάτι στο οποίο δεν εμπλεκόμεθα εμείς. Αυτό το οποίο μπορώ να πω είναι ότι προσπαθούμε να κατανοήσουμε το θέμα των ομάδων προστασίας από το επίπεδο των υπηρεσιών και προστασίας που παρέχουν ανασκάφος. Προσπαθούμε να κατανοήσουμε αυτή την προσέγγιση και υποστηρίζουμε το ότι μέχρι σήμερα σε σχέση με την, ε, το βαθμό επιτυχίας αυτών των δράσεων, αυτό το Σαββατοκύριακο υπήρξαν δύο επιδίων σκαφών που απετράπησαν λόγω προειδοποιητικών πυροβολισμών που ε, προήλθαν από αυτά τα σκάφη που εδέχονται ε, επιθέσεις. Πρέπει όμως να αναγνωρίσουμε ε, και να δεχθούμε ότι πρέπει η ναυτιλία να προστατεύεται επαρκώς. Προσπαθούμε με τα σκάφη τα οποία περιπολούν σε αυτή την περιοχή να διασφαλίσουμε ότι θα ε, ε, επιτυγχάνεται αυτός ο στόχος και βλέπουμε ότι είναι διαφορετικά τα αποτελέσματα σε σχέση με τις δράσεις. Όμως στον κόλπο του Άντεν και με την ε, αύξηση αυτών των περιστατικών πρέπει να δούμε ότι είναι μια πραγματική ανάγκη. Υπήρξαν ερωτήσεις όσον αφορά την διακυβέρνηση και την ασφάλεια. Θα μπορούσα εγώ ίσως να πω κάτι, αλλά από πλευρά ε, το, του συναδέλφου που ε, παρακολουθεί εκ του σύνεγγυ στα θέματα μπορούμε να αφήσουμε, μπορώ να αφήσω και να απαντήσει ο κύριος Ρόντος ε, για αυτό το θέμα ίσως. Και κάτι άλλο που είμαι βέβαιος ότι ο κύριος Ρόντος θα ήθελε να απαντήσει είναι το θέμα των νέων πειρατών και για τους νέους πειρατές όπως γνωρίζουμε και σε σχέση και με το οργανωμένο έγκλημα βλέπουμε ότι υπάρχει αυτή ε, αυτό το πρόβλημα και εναλλακτικές δυνατότητες πρέπει να αναζητηθούν ώστε να μπορέσουν να βρουν κάτι άλλο να ασχοληθούν πέρα από την πειρατεία. Στρεφόμενος στα θέματα που αναφέρθηκαν για το αν πρέπει να περνάμε στην ξηρά, στη στεριά με τις δράσεις μας και εδώ θα ήθελα να αναφέρω ότι η δική μου αποστολή ελέγχεται από την Επιτροπή Ασφάλειας ε, και Άμυνας. Έχω αυστηρούς κανόνες ε, για τις δράσεις μας και η δική μου αποστολή έχει επικεντρωθεί αυστηρά στην αντιμετώπιση πειρατείας και τρομοκρατίας. Και τα δύο είναι συμπτώματα ως φαινόμενα μιας ε, αποτυχημένης χώρας που βρίσκεται υπό Και εδώ φυσικά θα πρέπει να δούμε τι πρέπει να γίνει και με το πρότυπο το οποίο πρέπει να προαρθεί για να αντιμετωπιστεί αυτό το φαινόμενο. Σε σχέση με σχέσεις με άλλες χώρες συζητούμε με τους Κινέζους, υπάρχει με επιτυχία ένας θεσμός που ξεκίνησε κάποια χρόνια πριν που είναι το Shared Awareness and Deconfliction που δημιουργήθηκε από την NAFOR, CMF και το ΝΑΤΟ και σήμερα έχει πολλές συνιστώσεις και είχαμε στον Παχρέν μια συνάντηση πρόσφατα. Αυτά οδηγούν στο να συνέρχονται οι εμπλεκόμενοι της διεθνούς κοινότητας και αποδεικνύεται ότι είναι ένα αξιόλογο φόρουμ, ένα αξιόλογο μέσο για να έχουμε αυτές, αυτές τις επαφές ε, περιφερειακά. Όχι μόνο για να συζητούμε, αλλά για να σημειώνεται αυθεντική πρόοδος ε, στις δράσεις μας. Ε, και πρόσφατες επιτυχίες είναι ο μεγαλύτερος συγχρονισμός προστασίας νιοπομπών όσον αφορά αυτά τα ύδατα, αυτές τις περιοχές από πλευρά της διεθνούς κοινότητας. Και κάποιες συγκεκριμένες ερωτήσεις για την, Ινδία, την ε, ε, Σομάλιλαντ και τις πτυχές αυτές που συναρτώνται με τις ε, πολιτικές συνιστώσεις. Ίσως ο κύριος Ρόντος θα ήθελε να σχολιάσει περισσότερο αυτά. Συνεργαζόμαστε με την Ινδία υπό την πτυχή αυτού του διαλόγου θα υπήρχε η επιθυμία να υπάρχει ε, ένα ενιαίο πλαίσιο υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών ίσως. Όπως έχουν όμως τα πράγματα αυτή τη στιγμή επικοινωνούμε με τους Ινδούς, ε, έχουμε ανταλλαγή πληροφοριών και απόψεων, ιδιαίτερα όσον αφορά και την αντιμετώπιση ακριβώς των, της επιθέσεις που δέχονται τα σκάφη που ε, όσον αφορά την ε, Ινδική συνιστόσα θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η όλο και μεγαλύτερη συμμετοχή της Ινδίας στην απελευθέρωση ή της δράσης ε, κατά των πειρατών. Είχε αναλυφθεί τέτοια δράση για την ε, απελευθέρωση Ινδών, διασφαλίστηκε η απελευθέρωση πάνω από 45 Ινδών ναυτικών με αυτόν τον τρόπο. Νομίζω για την, ε, ε, το θέμα της παρέμβασης για την ε, ίδια τη Σομαλία και τι θα μπορούσε να γίνει. Πολύ δύσκολο να απαντηθεί. Παρακολουθούμε εκ του σύνεγγιστο τι συμβαίνει στη Σομαλία. Πάλι εδώ ο κύριος Ρόντος ίσως θα είναι ο πιο ενδεδειγμένος να τοποθετηθεί σε αυτό. Το επόμενο... Κάποιος χρησιμοποίησε την έκφραση military presence ashore, η στρατιωτική παρουσία στην ξηρά. Για να είμαστε σαφείς, ε, εδώ δεν είναι το θέμα της ε, στρατιωτικής παρουσίας στην ε, ξηρά υπό την ΝΑΦΟ, υπό τους όρους και προϋποθέσεις που έχουμε σήμερα απέναντί μας θα ήταν ίσως αντιπαραγωγική μια τέτοια παρουσία. Αυτό που έχουμε υπόψη σε σχέση με τις παράκτιες περιοχές είναι μια χειρουργικού χαρακτήρα δράση. Δηλαδή να υπάρξει η αντιμετώπιση στο χώρο που είναι υπό τον δικό μας έλεγχο, η αντιμετώπιση για παράδειγμα τέτοιων φαινομένων όσο όσον αφορά και την χρήση και ελικοπτέρων αεροπλάνων. Θέλουμε να το κάνουμε αυτό Αποκινούμε τους Σομαλούς και σε υποστήριξη των, από τους Σομαλούς. Αλλά πρέπει να το δούμε αυτό σε σχέση με την ατιμορρησία που απολαμβάνουν αυτή τη στιγμή οι πειρατές. Και αυτό είναι το κλειδί για αυτούς. Αν δεν έχουν αυτή την αυτονομία και ανεξαρτησία και ατιμορρησία δεν θα μπορούν να δρουν αυτόν τον τρόπο. Και το θέμα για την αλληλεία, η παρατήρηση, η εποπτεία της αλληλευτικής η δραστηριότητας ε, κατά το ξεκίνημα αυτής της δράσης ήδη είναι κάτι το οποίο ε, ε, καθημερινά κάνουμε. Γνωρίζουμε πολύ καλά πώς προσεγγίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση τα θέματα της παράνομης αλληλείας και των, της απόρριψης τοξικών αποβλήτων και πάντα πρέπει έτσι να τα αντιμετωπίζουμε και σε συνεργασία με τους Ομαλούς. Πολύ μικρής κλίμακας αλίας σε απόσταση 200 μιλίων από την ακτή της Σομαλίας ε, πατρίτες σήμερα και έχουμε στοιχεία που το ε, υποστηρίζουν αυτό. <clears throat> Σε σχέση όμως με την ε, ισχύ μιας αποκλειστικής οικονομικής ζώνης από πλευράς της Σομαλίας μέσα σε ένα τέτοιο πλαίσιο θα μπορούσε να συνεισφέρει να αποσαφινιστούν τα πράγματα όσον αφορά την αλληλεία και συναφείς δραστηριότητες. Έχουμε όμως αυτά τα ε, στοιχεία όσον αφορά ε, αυτές τις δραστηριότητες. Αυτές είναι οι σημειώσεις που είχα λάβει για τις ερωτήσεις σας και με βάση αυτές απάντησα. Αν κάτι δεν έχει απαντηθεί παρακαλώ να επανέλθετε ώστε να το απαντήσω μετά. Ε, Ο κύριος παρακαλώ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Μία ερώτηση και προς τους δύο προσκεκλημένους. Δεν υπάρχει κάποιος τρόπος να διακοπεί η ροή των χρημάτων, των ε, λίτρων που πληρώνονται. Γιατί αν δεν υπάρχει χρήμα τότε θα πάψει να υπάρχει και ο λόγος ε, για την πειρατεία. Και μία επιπλέον ερώτηση. Η Ρωσία συνεχίζει να εκτελεί τους ε, πειρατές. Ο τρόπος ε, ε, με τον οποίο τους σκότωναν είναι να τους εγκαταλείπουν σε πάρα πολύ μικρά σκάφη χωρίς νερό και φαγητό. Δεν ξέρω, μπορεί να μην το κάνουν ε, πια, αλλά να μην χρειάζεται να το κάνουν γιατί στάθηκε αποτελεσματικό. Κυρία Θα Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να συνδέσω το ερώτημα με την προηγούμενη ερώτηση. Βεβαίως εδώ συζητούνται κυρίως θετικά θέματα, αλλά θα ήθελα να αναφερθώ στις συνέπειες για το κράτος δικαίου. Στο Αμβούργο αυτή τη στιγμή γίνονται κάποιες δίκες κατά πειρατών και θα ήθελα να σας συστήσω να ρίξετε μια ματιά στο τι γίνεται σε αυτές τις δίκες. Τι είδους άνθρωποι είναι αυτοί οι οποίοι έχουν, για παράδειγμα, ε, συλληφθεί. Γιατί σε μεγάλο βαθμό πρόκειται για παιδιά. Παιδιά τα οποία συνελήφθησαν κάτω από συνθήκες που κανονικά ισχύουν μόνο για ενήλικες. Ε, και ε, ε, τελικά μετατρέπονται σε ενήλικες κάτω από μέσω αμφίβολων βιολογικών μεθόδων, βιολογιστικών μεθόδων. Δηλαδή ορισμένα από αυτά τα παιδιά δηλώνονται ότι είναι ενήλικες από ιατρούς και το παιδί αυτό παρέμεινε φυλακισμένο για μισό χρόνο παρόλο που δεν ήταν ενήλικο. Ε, θεωρώ ότι είναι πραγματικά φρικιαστικό αυτό το οποίο συμβαίνει με αυτούς τους ε, συλληφθέντες ε, πειρατές. Θα μπορούσαμε λοιπόν να δούμε τι τους άνθρωποι είναι και να εξάσουν και τα κίνητρά του. Ενδεχομένω, ορισμένοι πραγματικά αποφασίζουν αυτόβουλα να γίνουν μέλη αυτών των συμμοριών. Αλλά πολλές φορές είναι άνθρωποι που δεν το αποφασίζουν ε, ήδη. Ε, για παράδειγμα, συνθήκε στη Σομαλία όταν υπάρχουν περιχρωμένες οικογένειες, ε, κάποιο στον οποίο χρωστά τα χρήματα η οικογένεια, απαγάγει ένα από τα παιδιά αυτή τη οικογένεια και πολλές ε, φορές ε, λαμβάνονται αυτές οι αποφάσεις από ανάγκη. Για παράδειγμα ένα παιδί ή ένα αδελφός κάποιου ο οποίος έχει συλληφθεί ως πειρατής κλπ. Ε, νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να δούμε τι γίνεται. Θα ήταν μια εντατιγμένη λύση για να χειριστούμε την κατάσταση σε αυτή την πολύ κλονισμένη, βαθύτερα κλονισμένη χώρα. Ε, ίσως από ευρωπαϊκή πλευρά θα πρέπει να εξασφαλίσουμε τις ε, συνθήκες ε, ε, κράτους δικαίου όσον αφορά την παραμονή στις φυλακές και τις συνθήκες φυλάκισης των λεγόμενων πειρατών. Δηλαδή, κατά την άποψή μου, τα παιδιά αυτά τα οποία κατηγορούν για πειρατεία θα πρέπει να πάνε σε να κρατούνται σε αναμορφωτήρια ή σε ιδρύματα τα οποία προορίζονται για παιδιά. Okay. για Alex, um, Ευχαριστώ. ερωτήσεις πρώτα εκείνη για τους Ρώσους ε, και την θανατική ποινή. Δεν είναι δική μου δουλειά να σχολιάσω εγώ για πολιτικές άλλων κρατών, άλλων εθνών. Αυτό που θα μπορούσα να πω είναι ότι υπάρχουν πολλά ανεκδοτολογικά ή πολλές φήμες και ψήθυροι για το τι συμβαίνει ή όχι στη θάλασσα. Και σε σχέση με αυτό δεν είναι κάτι το οποίο έχει παρατηρηθεί υπό τους όρους ότι κάποιες χώρες ε, ε, συγκεκριμένων σκαφών, ε, τα σκάφη αυτά δεν υφίστανται επιθέσεις από κάποιους πειρατές. Είναι εγκληματίες αυτοί οι πειρατές. Προχωρούν στις περιοχές εκείνες όπου πιστεύουν ότι θα βρουν σκάφη και το πώς ε, μπορεί να δρουν κατά τους τελευταίους μήνες ε, για παράδειγμα σε σχέση με βοηθητικά βρετανικά σκάφη ε, από πλευράς αυτού του στόλου ή και ισπανικούς σκάφους της δικής μου δύναμης με πεζοναύτες στο ίδιο το σκάφος που αποτέλεσαν στόχους επιθέσεων δείχνει το τι συμβαίνει. Δεν υπάρχει περίπτωση βέβαια συνελήφθησαν αυτοί οι πειρατές. Τώρα για διακριτική αυτή μεταχείριση δεν είμαι βέβαιος αν υφίσταται και για την, ε, τα όσα συμβαίνουν όχι μόνο εγώ ο ίδιος αλλά και σε σχέση με όλα τα σκάφη, άνδρες και γυναίκες των δικών μας δυνάμεων, είναι ιδιαίτερα υπερήφανοι για το γεγονός ότι δρούν και λειτουργούν μέσα σε σαφώς καθορισμένα όρια όσον αφορά το διεθνές δίκαιο, την καταπολέμηση του εγκλήματος και το ανθρωπιστικό δίκαιο. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια διασφαλίζουμε ότι δρούμε, φυσικά με τους περιορισμούς που υπό τους οποίους δρούμε. Και μακροπρόθεσμα είναι ιδιαίτερα σημαντικό να βλέπουν ότι υπάρχει η λειτουργία και η δράση μας υπό αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις και περιορισμούς. στο τέλος τέλος θέλουμε να αλλάξουμε τα όσα συμβαίνουν στην ε, Σομαλία, να αλλάξει η άποψη των Σομαλών ε, έναντι της δικής μας δράσης, να δουν ότι είναι επικοδομητική η δράση αυτή και όχι απειλή ή επιβλαπτική για τους Σομαλούς. Για τα παιδιά έχετε απόλυτα δίκιο. Κάποια από τα που, τα φαινόμενα που βλέπουμε, βλέπουμε ότι υπάρχουν ανήλικοι και υπό τους όρους των δράσεών μας ε, για το αν μπορεί να δοθεί συνέχεια στην ε, ποινική δίωξη, αυτό μπορεί να γίνει μόνο όταν αυτοί παραδίδονται σε ένα ε, πλαίσιο ε, νομικής τάξης πραγμάτων όπου υφίστανται εχέγγυα για την ε, αντιμετώπιση τους ε, στην ποινική δίωξη περαιτέρω. Και θα έλεγα ότι αυτό εξαρτάται πάντα από το, την επάρκεια του δικαστικού και ποινικού συστήματος το οποίο διασφαλίζεται από τις αρχές τις οποίες παραδίδονται. Τώρα για τα όσα συμβαίνουν σε σχέση με τους Σομαλούς και τις δράσεις αυτές ε, είναι εκείνοι που βρίσκονται πίσω από αυτές τις δράσεις ως ε, ε, χρηματοδότες που πρέπει να καταπολεμηθούν. Και αν θέλουμε να καταπολεμήσουμε τη μάστιγα της πειρατείας που έχει πολλαπλές αρνητικές επιπτώσεις στην παγκόσμια ναυτιλία, το άμεσο κόστος όσον αφορά το, την ναυτιλία είναι δισεκατό, στο ύψος δισεκατομμυρίων δολαρίων ετήσια και έχει βαθύτατες επιπτώσεις σε όλη την περιοχή της Ανατολικής Αφρικής Αφρικής, ε, στις χώρες Ανατολικής Αφρικής. Αυτή η εγκληματική δράση που έχει τόσο σημαντικές επιπτώσεις πρέπει να αντιμετωπιστεί, αλλά φυσικά μέσα από τις ε, προϋποθέσεις και όρους και περιορισμούς υπό τους οποίους δρούμε. Ευχαριστώ. Bien, merci, ε, Ευχαριστούμε κύριε Νάβαρχε. Ο κύριος Ρόντους ήρθε και πραγματικά μόλις ήρθε από το κέρδος της Αφρικής ε, ακούσαμε μία κάποια εισαγωγή ε, είναι μια περιοχή που έχει όλο και πιο μεγάλη στρατηγική αξία για την Ευρώπη και ο διορισμός σας πραγματικά ανταποκρίνεται σε αυτό το ενδιαφέρον που επιδεικνύει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την ανάπτυξη της ασφάλειας αλλά και τις πολιτικές εξελίξεις στην περιοχή και από αυτή την άποψη η συνδιάσκεψη που έγινε στο Λονδίνο τέλη του μηνός Φεβρουαρίου σηματοδότησε μια σημαντική ε, φάση, ίσως όχι καθοριστική, αλλά πάντως ενδεικτική για την, πολιτική διαδικασία των πολιτικών εξελίξεων στη Σομαλία. Ίσως ε, βεβαίως ε, θα πρέπει να πούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ήταν ιδιαίτερος ε, παρούσα σε αυτή τη συνδιάσκεψη, έστω και αν συμμετείχε σε αυτήν η κυρία Άστον και εσείς ο ίδιος. Αλλά οι προσπάθειες που κάνει, που κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι επαρκής. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν ε, κάποια σημαντικά αποτελέσματα για τα οποία θα μπορούσατε να μας μιλήσετε και επίσης θα μπορούσατε να μας αξιολογήσετε τις πρόσφατες εξελίξεις στη Σομαλία, ε, τι γίνεται με την Αιθιοπία και την Κένια για παράδειγμα. Σας ευχαριστούμε που κάνατε ό,τι μπορούσατε για να έρθετε μαζί μας σήμερα το πρωί. Έχετε το λόγο. Uh, I'm very pleased to be Χαίρομαι που είμαι πάλι μαζί σας. Ζητώ συγγνώμη γιατί καθυστέρησα. Αλλά χθες στις 5 το απόγευμα ήμουν στο Μογκαντίσο. Και το μόνο που με καθυστέρησε για να έρθω εδώ ήταν η σειρά το ταξί που δεν υπήρχαν στο αεροδρόμιο των Βρυξελών. Είμαι βέβαιος ότι ο Ναύαρχος Πότς σας έδωσε ήδη ως συνήθως μια ιδιαίτερα πλήρη παρουσίαση. Λίγα πράγματα θα ήθελα να προσθέσω σε επίπεδο πολιτικό και να αναφερθώ γενικότερα στο πολιτικό πλαίσιο. Ίσως για να φανώ λίγο πόνηρος, να αναφερθώ σε δύο θέματα για την πειρατεία. τι μπορεί να συγκρίνει κανείς το παρελθόν με αυτό το οποίο συμβαίνει σήμερα. Είναι μια λύση που υπήρχε παλαιότερα. Η σταύρωση των πειρατών ήταν ένας τρόπος για την αντιμετώπιση τους ιδιαίτερος αποτελεσματικός. Ζούμε όμως σε μια διαφορετική εποχή. Και αυτό που ονομάζουμε ο χρυσός αιών της πειρατείας, δηλαδή ο 18ος αιώνας, όπου υπήρχαν τότε ορισμένοι Βρετανοί, κύριοι ιδιαίτερα γνωστοί. Ένας από αυτούς ήταν ο Τζον Έμπερι. Δεν ξέρω αν έχετε ακούσει γι' αυτόν. Ο Τζον Έμπερι αποφάσισε να γίνει πλούσιος, α, συλλαμβάνοντας τα μεγάλα εμπορικά πλοία που πήγαιναν από τον κόλπο της ε, Ινδίας προς ε, την Αφρική και είχε τη βάση του στη Σομαλία Είχε μάλιστα ε, καταλυστεύσει κάποιες περιοχές γύρω στο 1640 όπως τον Πάιτο. Η παρουσία της πειρατείας εκεί λοιπόν είναι παλαιά και οι μέθοδοι που ακολουθήθηκαν ήταν ιδιαίτερα αποτελεσματικές. Αλλά να περάσω λίγο τώρα στα σοβαρά και να περάσω στα ευρύτερα προβλήματα τα οποία έχει ήδη θέσει ο Πρόεδρός σας. Βρισκόμαστε σε μια φάση πλέον όπου είναι προφανή η βούληση της διεθνούς κοινότητας να αποτρέψουν τους Σομαλούς να εξάγουν την αστάθεια που αντιπροσωπεύουν στις οικονομίες μας και στις κοινωνίες μας. Αυτό είναι κάτι το οποίο λειτουργεί πράγματι αποτρεπτικά. Αυτά τα οποία συμβαίνουν μπροστά στις ακτές της Σομαλίας είναι κάτι το οποίο έχει συνεισφέρει σε ένα ευρύτερο πλαίσιο μέσα στο οποίο αυτοί οι οποίοι επιθυμούν να αποσταθεροποιούν τη Σομαλία αρχίζουν να συνειδητοποιούν ότι θα βρουν πλέον αντιπάλους απέναντί τους. Αντιπάλους οι οποίοι θα εμείνουν στην καταπολέμησή τους και θα περιορίσουν κατά πολύ την ικανότητά τους να αποσταθεροποιούν. Πέραν αυτού, να σας ε, ενημερώσω λίγο περισσότερο τους τελευταίους μήνες, όπως είπε ο Πρόεδρος, ε, ε, υπήρξε η διάσκεψη του Λονδίνου, υπήρξαν όμως και αρκετές εξελίξεις επιτόπου. Και εκεί θα ήθελα να στρέψω την προσοχή σας. Υπάρχουν τρεις βασικοί φορείς οι οποίοι εξελίσσονται παράλληλα και οι οποίοι θεωρητικά θα έπρεπε να είναι πιο συγχρονισμένοι και πιο συντονισμένοι για την παρέμβασή μας εκεί. Η ασφάλεια, η πολιτική κατάσταση και η ανθρωπιστική κατάσταση. Αυτό το οποίο έκανε η διάσκεψη του Λονδίνου είναι να υπογραμμίσει τη σημασία και των τριών αυτών παραγόντων και να υπογραμμίσει επίσης και την ανάγκη να υπάρξει βήμα προόδου και στα τρία αυτά θέματα. Για την ασφάλεια θα πω το εξής. Τα γεγονότα δείχνουν ότι η κατάσταση αλλάζει καθημερινά. Οι περισσότερες αλλαγές δεν είναι καν γνωστές. Η Σομαλία δεν συγκεντρώνει την προσοχή των μέσων ενημέρωσης καθημερινά, όμως υπάρχουν αλλαγές στη Σομαλία. Με το τελευταίο ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας που επιτρέπει την διεύρυνση και του μεγέθους και της εντολής της Αμτεσόκ, η οποία υποστηρίζεται και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, οικονομικά ενώ, ήδη διαπιστώνουμε ότι έχει ξεκινήσει ο προγραμματισμός και έχει σχεδόν ολοκληρωθεί για τη διεύρυνση της δράσης της αποστολής του ΟΗΕ και πέραν του Μογκαντήσου. Το Μογκαντήσου σήμερα έχει αλλάξει. Δεν είναι αυτό το οποίο ήταν εδώ και έξι μήνες. Δεν θα ήθελα να πω ότι εκεί θα πρέπει να πάτε για να περάσετε το Σαββατοκύριακό σας. Παρόλα αυτά είναι εκπληκτικό να βλέπει κανείς τη ζωή, την κίνηση, τα καταστήματα που ανοίγουν συνέχεια, τα σπίτια τα οποία ξαναχτίζονται, εφόσον οι ίδιοι οι Σομαλοί θέλουν να βάζουν τα χρήματά τους και να επενδύουν σε ένα μέρος σαν το Μογκαντήσου, αυτό κάνει τρομερή εντύπωση. Εγώ εξεπλάγιν. Ήδη με την αλλαγή που έχει επιτελεστεί μέσα και σε ένα μήνα, γιατί είχα πάει εκεί και πριν ένα μήνα. Ήδη η περιοχή η ελεγχόμενη έχει διευρυνθεί πάρα πολύ και υπάρχουν πολλοί οι οποίοι επιστρέφουν στα κτίρια, τα σπίτια από τα οποία είχαν διωχθεί πριν λίγο καιρό. Είχαν προσπαθήσει να ξεφύγουν ένα, δύο, πέντε, δέκα χρόνια. Και άλλοι πιστεύουν επίσης που ήταν στο Μογκαντήσου ότι μπορούν να επιστρέφουν σε άλλες περιοχές της χώρας. Και αυτό με φέρνει στο θέμα της ασφάλειας στην περιοχή. Συνειδητοποιείται ότι οι Αιθίωπες έκαναν μια εισβολή. Εκεί έχουμε συζητήσει επίσης ε, και τον ρόλο της Κένια. in ε, η Άμισομ έχει διευρυνθεί με δύο επιπλέον ε, μέλη, αλλά σε επίπεδο στρατιωτικό, από ό,τι φαίνεται, η Άμισομ δεν έχει προχωρήσει. Ο Σαμπάμπ εμένει και είναι πάντα κυρίαρχος. Οι Αιθίωπες έχουν φτάσει στην Παϊντόα και υπάρχουν και άλλες δράσεις οι οποίες εξελίσσονται και But what is this doing? If we are seeing a shift in the security, meaning who, who controls what, υπάρχει ανασφάλεια για το ποιος ελέγχει τι. Και αυτό είναι κάτι το οποίο μας οδηγεί στην πολιτική κατάσταση. Ποιος ελέγχει πολιτικά την χώρα. Και εδώ έρχεται ένας παράγων από αυτούς τους οποίους αναφέρθηκα πριν. Η πολιτική στη Σομαλία ορίζεται εν πολλής από τις επιθυμίες της διεθνούς κοινότητας. Και πολλοί Σομαλοί πιστεύουν ότι αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί. Δεν μπορεί η μεταβατική περίοδος να συνεχίζεται τόσο πολύ. Παρ' όλα αυτά, οι τοπικές διαπραγματεύσεις οι οποίες συνεχίζουν να εξελίσσονται έτσι ώστε να υπάρξει μια κάποια μορφή διοίκηση για να αντικαταστήσει αυτό το οποίο ελέγχει το Σαμπάμπι ή Σαμπάμπ αλλά μιλάω για την κεντρική ε, και ίσως βόρεια Σομαλία. Για την υπόλοιπη Σομαλία ίσως θα πρέπει να πούμε διαφορετικά τα πράγματα. Αλλά πάντως εκεί συμβαίνει κάτι το οποίο αποτελεί μια τεράστια πρόκληση. Γιατί οι στρατιωτικές δράσεις ε, ανοίγουν χώρο οι γυρεότεροι των φυλών, οι αρχηγοί των φυλών ζητούν περισσότερη βοήθεια και ζητούν περισσότερες διοικητικές δομές. Πρέπει λοιπόν να υπάρξει ένα συγχρονισμός ανάμεσα στην ασφάλεια και στην πολιτική. Εκεί και όπου κάποιες περιοχές ανακτώνται, πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα παροχής ασφάλειας στους κατοίκους της περιοχής έτσι ε, ώστε οι κοινότητες να δουν ότι έχει αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο ζουν, με τον οποίο οργανώνουν τη ζωή τους και νιώθουν ασφαλείς. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να έχουμε χρήματα στη διάθεσή μας για να προχωρήσουμε πάρα πολύ γρήγορα. Πρόκειται για μια παραδοσιακού τύπου πρόκληση, στην οποία θέλω να επιστήσω την προσοχή σας. Τίποτα δεν είναι χειρότερο από το να επενδύει κανείς τεράστια ποσά για να απελευθερώνει κομμάτια της χώρας και να βλέπει μετά ότι η ολοκλήρωση των περιοχών αυτών ε, σε επίπεδο ανθρώπινων πόρων έχει μείνει πίσω. Εγώ λοιπόν προσπαθώ να δω αυτή τη φάση πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε καλύτερο συντονισμό. Τώρα, για την ευρύτερη ε, πολιτική κατάσταση. Η διάσκεψη του Λονδίνου ενίσχυσε ή υπογράμμισε εκ νέου το γεγονός ότι τον Αύγουστο όπως είχε αποφασιστεί πέρυσι θα υπάρξει μια νέα πολιτική οργάνωση. Αυτό το οποίο συμβαίνει τώρα είναι ότι οι βασικοί ηγέτες συναντήθηκαν στην πρωτεύουσα του Πούντλαντ, δις θα συναντηθούν πάλι στις 25 Μαρτίου, στόχοι τους είναι να προσπαθήσουν να κάνουν μια πρόταση για το Σύνταγμα η οποία θα κατατεθεί σε μια συντακτική συνέλευση. Η συντακτική συνέλευση θα περιλαμβάνει περί τα χίλια άτομα. Θα επιλογούν με διαφορετικές μεθόδους και από την κυβέρνηση, θα υπάρχουν διαβουλεύσεις με τους παραδοσιακούς ηγέτες, και θα συμμετέχουν επίσης ε, και εκπρόσωποι των τεσσάρων μεγάλων φιλετικών ή εθνοτικών ομάδων συν ε, κάποιους ε, και συν τους υπόλοιπους των μικρότερων. Μέχρι τα μέσα Μαΐου θα έχει ήδη συγκληθεί η συνέλευση αυτή, θα έχει εγκρίνει όχι μόνο μία πρόταση συντάγματος, αλλά θα έχει εγκρίνει και τα ονόματα τα οποία θα πρέπει να πάρουν μέρος στο νέο κοινοβούλιο ε, το τελευταίο κοινοβούλιο, το μεταβατικό δεν ήταν ε, καρπός ε, εκλογής βέβαια. Γι' αυτό λοιπόν θα φτάσουμε, αν πάνε καλά τα πράγματα, τον Ιούλιο, τον Αύγουστο με ένα νέο κοινοβούλιο, το οποίο θα εκλέξει και θα επικυρώσει το νέο σύνταγμα, τη νέα κυβέρνηση και θα εκλέξει κυρίως ένα πρόεδρο. Τώρα αν θα είναι αυτός ή όχι θα δούμε. Αυτή είναι η διαδικασία όπως προβλέπετε. Όλοι ελπίζουν και όλοι επιμένουν ότι αυτά τα στάδια θα πρέπει μέχρι τον Αύγουστο να έχουν διανηθεί. Επιμελητιακά είναι δύσκολο αλλά εφικτό. Παρ' όλα αυτά όταν είπα αυτές τις μέρες, ε, όταν ήμουν στο Μογκαντήσο είχα συζητήσεις και όλοι προσπαθούν να το πετύχουν αυτό που είπα. Και θα ήθελα να περάσω τώρα πριν περάσω στο επόμενο θέμα, να θέσω δύο-τρία επιμέρους θέματα για, το, για τον καταστατικό χάρτη. Όλοι γνωρίζουν ότι δεν μπορούμε να έχουμε ένα τέλειο σύνταγμα το οποίο θα προταθεί σε χιλίους ανθρώπους που θα κληθούν να αποφασίσουν μέσα σε δύο εβδομάδες. Όχι, θα πρέπει να έχουμε ε, μία πρόταση περιληπτική η οποία θα περιλαμβάνει τις βασικές αρχές και η οποία τους επόμενους μήνες θα γίνει αντικείμενο εκλέπτυνσης και ανάλυσης. Και εδώ ερχόμαστε στο ομοσπονδιακό χαρακτήρα. Πόσο ομοσπονδιακός ή συνομοσπονδιακός θα πρέπει να είναι ο χαρακτήρας της χώρας. Ποιος θα είναι ο βαθμός της αυτονομίας και ποιος ο βαθμός της συγκέντρωσης. Παραμένει το θέμα του Σομάλιλαντ, το οποίο έχει ζητήσει διεθνή αναγνώριση, έχει αυτό ανακηρυχθεί ανεξάρτητο εδώ και αρκετό καιρό και νομίζω ότι όλοι στην Σομαλία συνειδητοποιούν πλήρως το ότι σήμερα θα πρέπει, τώρα πλέον θα πρέπει να υπάρξει μια κάποια συνταγματική ρύθμιση η οποία να αντιμετωπίζει και να αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα ότι πολλές περιοχές της Σομαλίας έχουν γίνει όλο και περισσότερο αυτόνομες. Χωρίς ε, να φτάσουμε στη φάση όπου θα πούμε ότι οι χώρες αυτές έχουν γίνει ανεξάρτητες ή όχι. και μπορεί ντε γιούρε να αποσκυρτήσει από την χώρα. Αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό είναι το θέμα. Είναι κάτι το οποίο είχαμε και ε, να αντιμετωπίσουμε στο παρελθόν και στην ε, εγγύς περιοχή μας, δηλαδή στα Βαλκάνια. Ένα άλλο θέμα είναι το φιλετικό θέμα. Η χώρα αυτή θα γίνει χώρα Σαρία ή όχι. Ανησυχούν οι γειτονικέ χώρες γιατί πιστεύουν ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να νομιμοποιήσει, θα έλεγα, την βίαιη επέκταση κάποιων θρησκευτικών πρακτικών και στις δικές τους γειτονικές χώρες. Υπάρχει δηλαδή και εξωτερική διάσταση. Τώρα, για την περιφερειακή πάντα διάσταση, να πω ότι ας μην έχουμε ψευδεστήσεις, δύο γειτονικές χώρες της Σομαλίας έκαναν μια απλή στρατηγική στρατιωτική επιλογή και είπαν ότι θα πάνε στη Σομαλία πριν εισβάλλει η Σομαλία σε αυτούς, για να το πω έτσι λίγο ξερά. Αυτοί που πιστεύουν ότι η αύξηση των προσφύγων, του αριθμού των προσφύγων, η αύξηση της τρομοκρατικής δραστηριότητας έφυγε και την Αιθιοπία και την Κένια και θεωρήθηκε ανυπόφορη η πίεση αυτή πλέον. Ιστορικά κάνει εντύπωση το ότι η Αφρικανική Ένωση ομόφωνα ε, υποστηρίζει ε, την αποστολή άμυσων. Αυτό είναι θα έλεγα πάρα πολύ σημαντικό και θεωρώ ότι είναι κάτι το καθοριστικό για τις σχέσεις που έχουμε για την Αφρική, ότι σε περιφερειακό επίπεδο δηλαδή υπήρξε το θάρρος να πάρουν μια τολμηρή απόφαση στρατιωτικά και να προσπαθήσουν να αποκαταστήσουν τη τάξη ε, της χώρας αυτής. Μιλάμε για μια περιοχή δηλαδή η οποία ανησυχεί για την ασφαλειά της και εγώ τους επόμενους μήνες θα έλεγα ότι μιας και έχουμε πετύχει εμείς τη δική μας ενεργασία και ολοκλήρωση σε επίπεδο ασφαλείας πρέπει να βοηθήσουμε και αυτούς. Τώρα να αναφερθώ στο λεγόμενο αναπτυξιακό σκέλος ή την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού. Θα ήθελα να πω ότι ανησυχώ γι' αυτό και γι' αυτό θα σας ζητήσω να πιστέψετε το ότι δεν μπορεί κανείς να απομονώσει την πολιτική από τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά της παρουσίας μας εκεί. Άλλο η πολιτική να πούμε δηλαδή, άλλο η ασφάλεια, άλλο η κοινωνική ανάπτυξη κτλ. Όχι. Μία είναι η πραγματικότητα. Υπάρχουν στρατιωτικές παρεμβάσεις, υπάρχουν πολιτικές παρεμβάσεις και πολιτικές διεργασίες που έχουν σαν στόχο την καλύτερη ζωή και υπάρχει επίσης ταυτόχρονα και η ανάγκη να υπάρχει καθαρό νερό, να υπάρχουν σχολεία, να υπάρχουν τα λεγόμενα κοινά αγαθά. Θεωρώ λοιπόν ότι σε αυτή τη φάση δεν έχουμε σε επίπεδο εξωτερικής παρέμβασης ολοκληρώσει την παρουσία μας σύμφωνα με τις ανάγκες των Σομαλών. Πρέπει να προσπαθήσουμε να εντοπίσουμε με σωστό τρόπο ότι εν πάση περιπτώσει έχει φτάσει η ώρα να δούμε στο σύνολό της την κατάσταση. Αλλάζουν τα θέματα στον τομέα της ασφάλειας, αλλάζουν τα θέματα στον τομέα της πολιτικής. Και πώς εσείς που είστε πολιτικοί ε, θα έλεγα πρωταγωνιστές δεν θα προσφέρετε στην περιοχή αυτή μόνο λόγια όμορφα αλλά συγκεκριμένη βοήθεια. Έφτασε η στιγμή τώρα να κάνουμε αυτό το οποίο θα χαρακτήριζα εγώ κάλυψη, πλήρη και πολλαπλή κάλυψη ε, των αναγκών μέσω των λεγόμενων πακέτων σταθεροποίησης. Και ασφάλεια από τη μία και πολιτική σταθερότητα από την άλλη και βοήθεια για την ανοικοδόμηση να νιώσει η κοινότητα αυτή της περιοχής ότι ε, πράγματι κάποιοι βοηθούν το θέμα είναι ότι πρέπει η παρέμβαση αυτή να γίνει σε εκατοντάδες περιοχές. Έχουμε όμως την ικανότητα να το κάνουμε. Έχουμε τα χρήματα για να το πετύχουμε. Αλλά για να το πετύχουμε πρέπει να συντονιστούμε. Έχουμε έξι μήνες με ένα χρόνο έτσι ώστε σε επίπεδο πολιτικό να ελέγξουμε την κατάσταση και να νιώσουν οι Σομαλοί ακόμα πιο πολύ ασφαλείς ακόμα πιο ε, πολύ ικανοί να προχωρήσουν ε, απομακρυνόμενοι από τα θέματα της βίας. Και σε αυτό αναφέρθηκε επίσης ε, και ο Ναύαρχος για την εκστρατεία εναντίον της πειρατείας. Δεν πρόκειται για μία απλή εκστρατεία. Υπάρχει μια συνολική αντίληψη η οποία λέει ότι οι ίδιες οι κοινότητες οι οποίες στοχεύονται για μια τέτοια δράση δεν είναι αλήθεια αυτό. Αυτό που είναι αλήθεια είναι ότι εκτός των κοινοτήτων θα πρέπει να στοχεύσουμε. Και ταυτόχρονα, όπως έλεγα και για άλλες περιοχές της Σομαλίας, η εκστρατεία σταθεροποίησης δίνει νέου τύπου κίνητρα στις κοινότητες αυτές. Οι ηγέτες λοιπόν των φυλών, οι νέοι, θα πρέπει να νιώθουν ότι μπορεί να έχουν ένα μέλλον, διότι η πειρατεία είναι ελκυστική βέβαια για αυτούς, αλλά τη στιγμή που θα βρεθούν στη φυλακή καταλαβαίνουν ότι δεν πάει πουθενά. Λοιπόν, έχουμε αρχίσει να παίρνουμε κάποια μηνύματα ότι οι σοφοί, θα έλεγα και οι ηγέτες των εθνοτικών ομάδων νιώθουν πλέον ότι αυτή η κατάσταση δεν πάει πουθενά. Το θέμα είναι όμως μας ρωτούν πώς θα μας βοηθήσετε να βγούμε από αυτό και δεν μπορούμε να πετύχουμε στην βοήθειά μας αν δεν ξεκαθαρίσουμε ότι η αποτροπή πρέπει να είναι ισχυρή και η αποτροπή πρέπει να είναι αποτελεσματική και σκληρή. Αν δεν νιώσουν την απειλή, τότε θα συνεχίσουμε να είμαστε μάρτυρες του προβλήματος. Και επανέρχομαι λοιπόν στο θέμα της πειρατείας. Ο τρόπος με τον οποίο θα αντιμετωπιστεί η πειρατεία είναι κάτι το οποίο δείχνει το τι συμβαίνει στην Σομαλία, θα καθορίσει το τι συμβαίνει στη Σομαλία και η καταπολέμηση της πειρατείας θα πλαισιώσει τη σταθεροποίηση της χώρας. Ιδιαίτερα μετά από αυτά τα οποία συμβαίνουν τους τελευταίους μήνες θεωρώ ότι τους επόμενους μήνες τα πράγματα μπορούν να πάνε καλά όχι μόνο προς δικό μας όφελος αλλά κυρίως των ιδίων των Σομαλών. Ευχαριστούμε πολύ για αυτή την παρέμβαση. Πριν δώσω το λόγο στους ε, συναδέλφους και συγχωρέσατε με που είμαι τόσο κοινότοπος, αλλά δεν έχουμε καθημερινά κάποιον που μόλις ήρθε από το Μογκαντήσου, όπως συμβαίνει σήμερα. Η πρώτη μου ερώτηση συνδέεται με αυτό που αποκαλέσατε ως αλλαγή, μετατόπιση της ασφάλειας, ε, security shift, σε σχέση με το ρόλο της ε, Αμισόμ και τις ε, συνδρομή των άλλων χωρών. Ε, στην ίδια τη Σομαλία, πώς σκέφτεσαι ότι οι ίδιοι Σομαλοί βιώνουν αυτή την αλλαγή, στα, την καμπή στα θέματα ασφάλειας. Δηλαδή η αμισόμη γίνεται αποδεκτή, τα ξένα στρατεύματα γίνονται αποδεκτά, γιατί τέλος αυτή η αλλαγή μοντέλου όσον αφορά την ασφάλεια έχει συμβεί επιτελεστή και στο παρελθόν και πολύ γρήγορα τα ξένα στρατεύματα στην Αιθιοπία δεν έγιναν αποδεκτά και τελικά ενίσχυσαν την Σαμπάμπ. Ε, μήπως θα καταλήξουμε λοιπόν σε αυτό το σημείο, δεν είμαστε βεβαίως ακόμα εδώ, αλλά ίσως εγκυμονείται αυτός ο κίνδυνος. Και πώς θα μπορούσαμε να διαχειριστούμε αυτό το κίνδυνο σε ένα άστιμο, ε, διάστημα. Ο κύριος Γκάλετ ε, θέλει να πάρει το λόγο. Ναι, μια ερώτηση που αφορά την ε, περιοχή αυτή στην οποία αναφερθήκατε, τον τομέα αυτό στον οποίο αναφερθήκατε. Είπατε ότι με τη διεύρυνση της εντολής και, την, ε, τους, ε, και τους από την Κένια, η Άμισόμ, είναι ενεργή και σε αυτή την περιοχή του Μογκατήσου και την νότια περιοχή. Αν δούμε το χάρτη, Έχουμε το Σομάλιλαντ, το Πούντλαντ δυτικά και ανάμεσα υπάρχει μια ελεύθερη περιοχή όπου θεωρητικά τουλάχιστον θα μπορούσαν να παραμείνουν αυτές οι πολιτοφυλακές και που ενδεχομένως θα μπορούσαν να λειτουργήσουν σαν μια βάση για τους πειρατές. Ε, θα μπορούσαμε ίσως να συνδέσουμε αυτές τις δύο αποστολές, την Αμισόμ και την Αταλάντα, ίσως αυτές οι δύο θα ήταν κάποτε σε θέση να καλύψουν αυτό το κενό που υπάρχει εδώ. Γιατί αυτό το οποίο γίνεται τώρα στο Μογκαντήσου, αυτό το οποίο κάνουν οι αρχηγοί των φυλών, ε, ή το επιθυμούν μάλλον, να υπάρξει μια βελτίωση στη δίκηση, ίσως να μπορεί να γίνει ε, σε όλη τη χώρα. Για ποια χρονικά διαστήματα μιλάμε τώρα, όταν λέτε, αναφέρεστε στον Αύγουστο, λέτε ότι θα ε, ε, υπάρξει μια καταστατική συνέλευση λοιπά, θα ψηφιστεί σύνταγμα. Μπορεί να υπάρξει αυτή η γεωγραφική επέκταση και σε άλλες περιοχές αυτών των διαδικασιών. Ποιες είναι οι δικές σας προσδοκίες από τη μία πλευρά τι μπορεί να αναμένει κανείς ε, ρεαλιστικά όσον αφορά την ε, ύπαρξη μιας πολιτικής βούλησης της Βρυξέλλης προκειμένου να συμμετάσχουν όλες οι χώρες μέλη εδώ. Ευχαριστούμε πολύ. Κυρία Νικολά έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Ε, ακολουθώντας όσα είπατε για την πειρατεία και το ιστορικό, μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι η Σομαλία ήταν πόλος ε, έλξης, ακόμα και στο 18ο αιώνα και τώρα. Για μένα αυτό το θέμα της πειρατείας είναι ένα θέμα που εμπίπτει στο οργανωμένο έγκλημα. Πιστεύω ότι δεν αφορά μόνο την κατάσταση των φτωχών Σομαλών, των παιδιών ή ενηλίκων, αλλά επίσης είναι ένα θέμα, ένα ζήτημα οργανωμένου εγκλήματος όπου υπάρχουν πολλές διεθνείς συνδέσεις. Ε, υπάρχει κάποια σχετική έρευνα. Έχουν ε, γίνει έρευνες, υπάρχουν πληροφορίες, γιατί είμαι σίγουρη ότι θα, υπάρχουν κάποιες σχετικές πληροφορίες. Ε, αλλά υπάρχει κάποιο κίνητρο να γίνουν αυτές οι έρευνες, γιατί τα ωφέλη για την πειρατεία δεν αφορούν μόνο τους Σομαλούς, αλλά και άλλους στη διάσκεψη του Λονδίνου λήφθη απόφαση να λήξει η εντολή της ε, προσωρινής, ε, ε, του προσωρινού θεσμικού οργάνου, του μεταβατικού θεσμικού οργάνου. Ε, πιστεύετε στη βιωσιμότητα της χώρας αυτής. Μιλάτε για μια ομοσπονδιακή προσέγγιση. Νομίζω ότι το Σομάλι Λαντ και η Πούντ Λαντ θα ε, ε, πρέπει να αποκτήσουν μια δυνατότητα να γίνουν βιώσιμες ε, περιοχές. Εάν έχουμε μια αποτυχία φέτος αυτή την προσέγγιση, νομίζω ότι αυτό θα είναι ένας μεγάλος κίνδυνος, γιατί μπορεί να κλιμακωθεί η κατάσταση. Αν δούμε ποιο είναι το πολιτικό πλαίσιο, το πολιτικό περιβάλλον, και, γειτον, και τι γίνεται στις γειτονικές χώρες. Νομίζω ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε να έχουμε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση. Αλλά το πραγματικό πρόβλημα αφορά το είδους της, τη μορφή της, που θα πρέπει να προσλάβει η χώρα στην οποία θα προσφέρουμε αυτή την ολοκληρωμένη προσέγγιση. Σε ποιους ακριβώς θα απευθύνεστε. Ευχαριστούμε πολύ. Ε, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αναφέρατε σύντομα ότι η υπάρχει αυτή η εξ, μείωση των Al-Shabaab αλλά μπορεί να επανεπιτεθούν. Αυτό τι σημαίνει, ότι μπορεί να επιτευχθεί μια συμφωνία μαζί τους σε διαπραγματεύσεις για την ειρήνη ή ένα συμβιβασμό. Υπάρχουν καθοδόν προσπάθειες για κάτι τέτοιο ή όχι. Δεύτερη ερώτηση, πέρυσι ο ειδικό ε, σύμβουλο Jack Lang για τα θέματα πειρατεία υπέβαλε προτάσει στο Συμβούλιο Ασφαλεία των Ηνωμένων Εθνών για την αντιμετώπιση των θεμάτων τη πειρατεία ε, με βάση την προσέγγιση τη ε, προσαγωγή στη δικαιοσύνη των υπεύθυνων τέτοιων εγκλημάτων. Έτσι θα έπρεπε να προχωρήσουμε. Τι θα έπρεπε από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Ένωση να υιοθετηθούν κάποιε από αυτέ τι προτάσει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ ευχαριστώ κύριο Στένοκ. Ευχαριστώ Κύριε Ρόντο, αναφέρατε ότι κάπως ε, κατακαιρματίζεται η διεθνής κοινότητα σε σχέση με την ε, προσέγγιση κατά πολέμησης της πειρατείας. Έχουμε την ε, ΝΑΦΟ, την Αταλάντη. Αυτό είναι ισχυρό επιχείρημα για την δράση υποπλευράς Ηνωμένων Εθνών στρατιωτικά και με την Amazon, Amazon και σε σχέση με τη συνιστόσα της Αφρικανικής Ένωσης. Είναι ρόλος για τα Ηνωμένα Έθνη. Πώς θα μπορούσε μια τέτοια προσέγγιση να υιοθετηθεί αποτελεσματικά. Και μια κυρία πίσω από μένα ανέφερε τα παιδιά από και 14 ετών και φυσικά σε σχέση με, την εγκληματική, ε, με εγκληματικές πράξεις μπορούν να θεωρηθούν ε, υπεύθυνα τέτοιου είδους άτομα πώς μπορεί να προσεγγιστεί το θέμα της ε, ευθύνης. Ε, ε, στη χώρα μας ένας 14χρονος για την διάπραξη σοβαρού εγκλήματος θα μπορούσε να καταδικαστεί. Πώς θα μπορούσε αυτό γενικότερα ίσως να εισαχθεί και σε σχέση με τα τεκμήρια για το ότι κάποια από τα χρήματα των ε, ε, πειρατικών αυτών πράξεων χρηματοδοτούν τις δράσεις των αντατών Σαμπάμ. Έχουμε κάποιες ε, αποδείξεις, κάποια αποδεικτικά στοιχεία. Υπάρχουν όλο και πιο στενές σχέσεις των Σαλαφιστών, των Αλκαϊντιστών και στην Αλκάιντα του Μαγκρέμπ και των άλλων Σαλαφιστών με την δυνατότητα να χρηματοδοτούνται από αυτά τα λίτρα Σαλαφιστές και ακραίοι τζιχαντιστές. Ε, ενδιαφέρομαι ιδιαίτερα για το θέμα της Σομάλιλαντ ε, και της ε, αναγνώρισης. Ιδιαίτερα ενδιαφέρομαι επειδή υπάρχουν άτομα από τη Σομάλιλαντ στη δική μου εκλογική περιφέρεια και ήταν και κτήμα, ήταν απικία της Μεγάλης Βρετανίας και έτσι σε σχέση με μια μη ικανοποιητική λύση που θα δυσαρεστούσε την Σομάλιλαντ δεν θα έπρεπε να την δεχτούμε πώς θα μπορούσαν να ικανοποιηθούν ε, οι απόψεις ε, των εκπροσώπων της Σομάλιλαν. Είχαν αποστείλει μια αντιπροσωπή στο Λονδίνο και ήταν ε, θετικό το ότι υπήρχε αυτή η παρουσία στο Λονδίνο. Μπορούμε να ξεπεράσουμε αυτό το πλαίσιο και να συμμετάσχουν στη συνταγματική τάξη πραγμάτων οι εκπρόσωποι της Σομάλιλαν. Θεωρούν ότι είναι ανεξάρτητο κράτος και αυτό θα μπορούσε να είναι ένα θετικό στοιχείο για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, της πειρατείας, τη διεξαγωγή δημοκρατικών εκλογών κτλ. Εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά τα κράτη-μέλη υπάρχει πολλές φορές η κατηγορία για τα δύο μέτρα και δύο σταθμά ή για ένα μικρό χρονικό διάστημα η Σομάλι Λάντε για την αναγνώριση που ε, θέλει να ε, πετύχει είναι να μπορέσει να θεωρείται μια χώρα ε, ανεξάρτητη υπό τα σύνορα τα οποία είχε στο παρελθόν. Πρέπει να είμαστε συνεκτικοί και συνεπείς και ε, να μην υιοθετούμε δύο μέτρα και σταθμά. Ούτως έχουν τα πράγματα. Αυτές είναι οι δικές μου ερωτήσεις προς τον κύριο Ρόντο. Ευχαριστώ. Merci, enfin, monsieur Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος ε, Λίζεκ έχει το λόγο. Ναι, e, για να είμαι ειλικρινής, όταν συζητούμε με κάποιον ο οποίος εκπροσωπεί την Ευρωπαϊκή Ένωση σε όλες τις γωνιές του κόσμου, λέμε πάντοτε ότι υπάρχουν, υπάρχει η συχνότητα των μέσων. Με εντυπωσιάζει το ότι είπατε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επαρκή μέσα όσον αφορά την περιοχή αυτή για την εκδίπλωση των δραστηριοτήτων. Επαρκή ως προς προς να παράξει τι. Αυτό είναι το πρώτο. Και δεύτερον, ποιο είναι ο ρόλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με τα μέσα αυτά τα οποία έχει στη διάθεσή τη η Ευρωπαϊκή Κοινότητα και ποιο ε, συμβάλλει στα μέσα αυτά για, τις, ε, για την επίτευξη αυτών των ε, δραστηριοτήτων. Ευχαριστούμε πολύ ο κύριος Κύρλοφ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Μια πολύ σύντομη ερώτηση. Εγώ θυμάμαι πολύ καλά αυτή τη λαμπρή επιχείρηση όταν ε, εξαφανίστηκαν οι τρεις ε, πειρατές ε, κατ' ουσία. Ποιο είναι, στις ΗΠΑ, ποιο είναι, ποιο είναι το ποσοστό των Αμερικανικών πλοίων που γίνονται αντικείμενο επιθέσεων. Βεβαίως κατανοώ ότι εμείς δεν έχουμε τις ίδιες ικανότητες όπως και οι Αμερικανοί. Αλλά αυτό είναι ένα παράδειγμα για το πώς θα μπορούσαν να μειωθούν όλες αυτές οι δραστηριότητες των πειρατών. Ευχαριστούμε πολύ. Δεν ξέρω αν δεν υπάρχουν άλλες παρεμβάσεις. Ίσως ο κύριος Ράντος να απαντήσει. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ας ξεκινήσω. Θα ξεκινήσω, θα λέγαμε το πιο κέριο ερώτημα το οποίο διατυπώσατε, Πρόεδρε. Και αν κατάλαβα σωστά την ερώτησή σας, θα ήθελα με τη δική μου διατύπωση να απαντήσω, με τα δικά μου λόγια. Αν ε, εσόν θα είχε τον κίνδυνο που θα αντιμετώπιζε αντί να είναι ένας ε, ειρηνοποιός ε, να θεωρηθεί ότι παρεμβαίνει και δημιουργείται μια αστάθεια. Εκείνο το οποίο με ενθαρρύνει είναι ότι έχουμε και τους ίδιους τους υπεύθυνους και είναι εκείνοι οι οποίοι λένε ότι μας δόθηκε η εντολή να εκαθαρίσουμε κάτι. Πού βρίσκονται όλοι οι άλλοι εμπλεκόμενοι για να παγιωθεί η κοινωνική συνιστόσα, η πολιτική, η οικονομική συνιστόσα. Οι, Αιθίω, οι Αιθίωπες έμαθαν το μάθημά τους, πιστεύω, από την τελευταία φορά. Είναι σαφές ότι ήταν απόλυτα σαφή, σαφής η πρόθεση να μπορέσουν να αποχωρήσουν. Δεν θέλουν και ε, όσον αφορά την ε, ΝΤΟΑ και τις ε, άλλες δράσεις για τη διασφάλιση της επικράτειας. Είπαν όμως κατά τα μέσα Απριλίου θα αποχωρήσουν και θα, είναι, θα έχουν εγκαταλείψει την περιοχή. Και σε σχέση με τα όσα συνέβησαν την τελευταία φορά, αυτό πρέπει να δούμε. Παρόμοια αναμένουν να πάρουν κάποιες, να δοθούν κάποιες πρόσθετες ε, δυνάμεις ε, ώστε να μπορέσουν να αντικατασταθούν οι αιθιοπικές δυνάμεις ε, στην περιοχή από την οποία θα αποχωρήσουν. Και αυτό δείχνει το τι εννοούσα με τη χαρτογράφηση όταν είπα ότι πρέπει να χαρτογραφήσουμε όλα αυτά. Πρέπει να τα μεταφράσουμε με πρακτικούς όρους ε, και ε, συνιστώσεις. Ε, τι θα πρέπει και τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να βοηθήσει με όλα τα κονδύλια τα οποία έχουν δοθεί. Θα θέλαμε οι επενδύσεις μας να στεφθούν με επιτυχία, να έχουμε ένα θετικό αποτέλεσμα. Πολιτικά να υπάρχει ένα θετικό αποτέλεσμα. Αυτό είναι το επίπεδο στο οποίο πρέπει να το δούμε. Αυτή είναι η πρώτη απάντηση. Τώρα, σε σχέση με τα κενά ή τα χάσματα τα οποία θα μπορούσαν να δημιουργηθούν, να προκληθούν με την Αταλάντη, κάνοντας η Αταλάντη το δικό της έργο, η Amazon το δικό της έργο, με τις ροές ε, που υπάρχουν, ποιος ελέγχει τι επιτόπου, το κενό που θα μπορούσε να προκληθεί. Και είμαι πεισμένος ότι βρισκόμαστε σε μια ε, δυναμικά εξελισσόμενη κατάσταση, ενρευστό, και τις τελευταίες ε, ημέρες ομιλώντας με τους ε, επικεφαλείς της ε, Amazon και οποιοδήποτε στρατιωτικά υπεύθυνος θα σας πει τη στιγμή που ξεκινά η στρατιωτική δράση όταν όταν προχωρεί, ε, προχωρά αυτή η δράση πρέπει να αντιμετωπίσει κανείς την πραγματικότητα που διαμορφώνεται και τις ευκαιρίες ε, και τους στόχους ε, που πρέπει να λαμβάνονται πάντα υπόψη προσαρμοζόμενοι πάντα στην πραγματικότητα. Θα δημιουργηθούν τώρα κάποια κενά, κάποια, κάποια, κάποια χάσματα. Η ολοκλήρωση αυτών των δράσεων θα πρέπει να ακολουθηθεί από άλλες δράσεις στο πολιτικό επίπεδο, αναπτυξιακό επίπεδο, ε, στο, επίπεδο ανθρωπιστικής βοήθειας. Ανθρωπιστικά λοιπόν θα πρέπει με σαφήνεια να δούμε αυτή τη συνιστόση Αν υπάρξει χώρος και δυνατότητα περιθώριο που μπορεί να αναπτυχθεί θα πρέπει η διεθνής κοινότητα να δραχθεί της ευκαιρίας και να το καλύψει με τις ανθρωπιστικές δράσεις ε, δρατώμενη της ευκαιρίας και ε, ε, στο ύψος των περιστάσεων με τις δράσεις που θα αναλάβει. Η ευκαιρία λοιπόν προσφέρεται να γίνει αυτό και δεν μπορούμε να τη χάσουμε αυτή την ευκαιρία. Τώρα, αν θα υπάρχει από πλευρά τη διοίκηση ε, των Σομαλών, αν θα υπάρξουν κενά ή όχι, μια και, θέλουμε, και κάποιοι θέλουν να, να γίνουν μέρο μια ε, κυβέρνηση, ε, όταν ε, κάποιοι επιτόπου φύλαρχοι ε, συγκρούονται. Ε, αυτό δεν είναι κάτι το ευταίο. Εκείνο το οποίο ελπίζω είναι ότι θα μπορέσουμε να έχουμε κανονικής πολιτικής ζωής διαδικασίες και διεργασίες ώστε όταν υπάρχουν τέτοιες διαφορές να επιλύονται στο πολιτικό επίπεδο και όχι με αλληλοσκοτομούς να προχωρεί η αντιπαράθεση. Τώρα, μεταβατική περίοδος, μετάβαση όσον αφορά και τον Αύγουστο. Ε, προσεγγίζοντας αυτό θα ήθελα να μας προβληματίσουν αυτά τα στοιχεία. Να μην κάνουμε το τέλειο, τον απόλυτο εχθρό του καλού, γιατί τότε δεν θα μπορέσουμε να έχουμε θετικά αποτελέσματα. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι θέτουμε στόχους, στοχοθετούμε και όταν θέτουμε κάποιους στόχους επικεντρωνόμαστε σε αυτούς για την επίτευξή τους. Αυτό είναι αυτό που πρέπει να κάνουμε. Περνάμε απο, περνώντας από φάση σε φάση και ε, υλοποιώντας τα διάφορα βήματα που πρέπει να κάνουμε στη Σομαλία δεν θα έχουμε μια τελειότητα, ένα τελικό τέλειο προϊόν ως αποτέλεσμα. Αυτό που πρέπει να προσπαθήσουμε να πετύχουμε είναι να υπάρξει μια συμφωνία γύρω από ένα πολιτικό πλαίσιο ως ε, πλαίσιο που θα δώσει τη δυνατότητα στους Σομαλούς να προχωρήσουν και να πούν έχουμε τώρα ένα πολιτικό σύστημα σε ένα ευρύτερο πλαίσιο που θα δώσει τη δυνατότητα πολιτικής στα από πλευρά μας μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Η αδιάκριτη χρήση των όπλων, δηλαδή η απεριόριστη αδιάκριτη ε, βία θα τιμωρείται και θα πρέπει άμεσα να αντιμετωπίσετε. Αυτό τι σημαίνει. Δημιουργία σομαλικού στρατού και σομαλικής αστυνομίας ε, που είναι αναγκαία ε, ως συνιστός. Δηλαδή η άσκηση του θεσμικού δυναμικού που πρέπει να διασφαλίσει το κράτος δικαίου, την ένωμη τάξη στην ε, Σομαλία. Για να προχωρήσουμε πρέπει να διασφαλιστούν αυτές οι συνιστώσεις. Στην Κωνσταντινούπολη διάσκεψη η Τουρκία θέλει να στεφτεί με επιτυχία διάσκεψη της ε, Κωνσταντινούπολης να υπάρξει ε, σε σχέση με τη συνταγματική ε, διάσκεψη τη συμφωνία για το Σύνταγμα, επιλογή μελών της, ε, του Κοινοβουλίου, της συνέλευσης και προϋποθέσεις που θα δημιουργηθούν για τις επόμενες φάσεις. Εκλογές, τώρα εκλογές πέρα από τον πρόεδρο της Βουλής δεν φαίνεται να είναι πιθανές αυτή τη στιγμή. Τώρα για το ότι τον Αύγουστο το ότι θα μπορούσαμε να τα καταφέρουμε καταφέρουμε αυτά, αυτή είναι μία φάση μόνο στην παγίωση, στην εμπέδωση της σταθερότητας στη Σομαλία και τη διασφάλιση της ασφάλειας των ατόμων, των πολιτών της ε, ε, Σομαλίας. Υπό αυτό το πρίσμα πρέπει να τα προσεγγίσουμε. Τώρα για την πειρατεία και το οργανωμένο έγκλημα Έχετε δίκιο, απόλυτα. Είναι οργανωμένο έγκλημα και πειρατέ, είναι εγκληματίε, είναι βέβαιο. Και λυπούμε πολύ για τα παιδιά τα οποία αποτελούν θύματα αυτή τη διεργασία και συμμετέχουν σε αυτό το εγκληματικό πλαίσιο. Είναι η χαμένη γενεά αυτή που ε, έχει ε, παρασυρθεί, α το πω έτσι, και εμπλέκεται μέσα σε ένα τέτοιο φαύλο κύκλο και πληρώνουν το αντίτιμο με την τιμωρία και την, ε, τις κυρώσεις ε, που ε, αυτά θα πρέπει να συνεπάγονται. Και απόλυτα σαφής είναι η τοποθέτησή μου και η άποψή μου. Αν σιγά σιγά σταδιακά περάσει αυτό το μήνυμα στις κοινότητες στην κοινωνία και αυτό ήσυχα με ήσυχο ήρεμο τρόπο θα πρέπει να προχωρήσει και να πιστούν οι γονείς και οι ενήλικες ότι αν θέλουν τα παιδιά τους να προστατευθούν. Αν θέλουν οι νέοι να προστατευθούν από το πεπρωμένο ενός ε, εγκληματία πειρατή νέου που έχει συλληφθεί και πρόκειται να προσαχθεί στη δικαιοσύνη και να τιμωρηθεί, τότε θα είναι σαφές ότι για τέτοια παιδιά αν ε, κάποιος ε, θα τα ή θα θέλει να τα οδηγήσει στην πειρατεία, δεν είμαι βέβαιος τώρα ότι μπορούμε να αναλύσουμε όλα αυτά τα στοιχεία για κάθε τέτοια περίπτωση, αλλά η παρατήρηση που έγινε κατέστησε σαφές αυτό το θέμα και είναι σαφές ότι είναι σημαντικό και το θέμα των φυλακών, αλλά πρέπει να δούμε τα πράγματα με τη σειρά. Το πιο σημαντικό που έχουμε μπροστά μας αυτή τη στιγμή ως προτεραιότητα και να το αναδιατυπώσω αυτό. Το να χτίζουμε φυλακές απλά και μόνο για να φυλακίζουμε, πειρα... Ε, φυλακές για να ε, φυλακίζουμε πειρατές ε, όπου υπάρχει η πιο φρικτή ε, μοίρα των ε, πολιτών από την ε, ε, άκρατη και αδιάκριτη βία η θεραπεία είναι το κράτος δικαίου και η ένομη τάξη. Αν θέλουμε ένομη τάξη και κράτος δικαίου στη Σομαλία πρέπει να δημιουργήσουμε το δικαστικό, πρέπει να δημιουργήσουμε τα σώματα ασφαλείας, την αστυνομία, την δυνατότητα σωστής προσαγωγής στη δικαιοσύνη και φυλάκισης. Και το θέμα των βιασμών Α Ας ε, ε, συλληφθούν λοιπόν ε, οι δράστες, υπάρχουν άλλοι που λαιλατούν, ληστές που λαιλατούν και κλέβουν. Όλες αυτές οι μορφές βίας, η ένομη τάξη και το κράτος δικαίου όλα αυτά συνεπάγονται. Δηλαδή ένα πλαίσιο που θα οδηγεί στην αποκατάσταση της δικαιοσύνης. Τώρα, για το άλλο, υπάρχουν ήδη τώρα διακριβωτικές και ανακριτικές ε, δράσεις και πραγματικά εντείνονται και σαν συνέπεια όλων των αποτρεπτικών δράσεων, ας είναι αυτό σαφές, όλοι όσοι θα συλλαμβάνονται θα είναι μια πηγή για πληροφορίες ε, και θα δείχνουν τι μπορεί να συμβεί με την σωστή και αποτελεσματική δίωξη και καταδίκη των υπεύθυνων. Γι' αυτό αυτά τα οποία συμβαίνουν είναι τόσο σημαντικά ως υποδειγματικά στην ε, δράση μας γνωρίζετε ότι δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν κάποια έκτακτα δικαστήρια απλά και μόνο επειδή υπάρχει το φαινόμενο της πειρατείας. Θα πρέπει να υπάρχει ένωμη τάξη, ε, μια δικαστική εξουσία η οποία θα δίνει συνέχεια με τις ανακρίσεις και τη διακρίβωση για την δίωξη και πάταξη της πειρατείας. Είναι απόλυτα λοιπόν σαφές ότι υπάρχει πρόοδος ε, από την άλλη πλευρά που σημειώνεται με αυτές τις ε, δράσεις ε, και τις ανακρίσεις και πρέπει να ενταθούν και να προχωρήσουν ακόμα περισσότερο. Τώρα κάποιος ανέφερε το θέμα ότι πιθανώς ε, οι οι αντάτες και οι πειρατές ε, συνδέονται ε, πέρα από το ιδεολογικό πεδίο χρηματοδοτικά με, τις, με τα λίτρα που εισπράττονται και την χρηματοδότηση που διασφαλίζεται. Αν λοιπόν οι σαμπάμπ, οι αντάρτες και οι πειρατές είναι ενδείξεις, συμπτώματα μιας διαλυμένης χώρας, είναι σαφές ότι οι μεν θα γνωρίζουν για την ύπαρξη των δε και θα συνεργάζονται. Τώρα, κατά πόσο συνεργάζονται αυτά εξαρτώνται όλα από τις συνθήκες και προϋποθέσεις επιτόπου. Είναι πιθανό να συμβαίνει αυτό. Είναι πολύ δύσκολο να εξευρεθούν τα τεκμήρια, αλλά αν τώρα οι Σαμπάμπα εξάγουν τα ε, κονδύλια αυτά, τότε είναι ποιο είναι εκείνο ο οποίο διαχειρίζεται αυτή την εξαγωγή κεφαλαίων, την οικονομική αυτή δράση. Και εδώ περνάμε τώρα στο επίπεδο τη ε, συνιστόσα αυτή στην ίδια τη Σομαλία και είναι μια ξεχωριστή συζήτηση. δεν έχω καμιά αμφιβολία ότι υπάρχουν συμφέροντα. Συμφέροντα τα οποία ε, το ένα με το άλλο συνεργάζονται και αυτά όλα μεταφράζονται μέσα σε ένα πλαίσιο των ε, πολιτικών διεργασιών της ίδιας Σομαλίας. Πρέπει λοιπόν σε αυτό να στραφούμε. Αυτά τα οποία είναι ενδείξεις και συμπτώματα του οργανωμένου εγκλήματος να μην έχουν την ευκαιρία να μεταφραστούν ή να μετουσιωθούν σε κάτι άλλο που θα είναι πάλι δίκτυο του οργανωμένου εγκλήματος όμως ε, που θα είναι σε ένα τελείως διαφορετικό πλαίσιο. Εμείς θα πρέπει λοιπόν να ακολουθήσουμε και να διώξουμε αυτές τις δράσεις. Είναι η επόμενη φάση της πρόκλησης που, στην οποία πρέπει να αποδηθούμε στην καταπολέμηση αυτών των φαινομένων. Τώρα για την ερώτηση που έγινε για το θέμα Al-Shabaab. Θέλω να είμαι προσεκτικός ώστε να μην υπάρξει παρερμηνία. Όταν λέω ότι συρρυκνώνονται οι ε, έχει υπάρξει μια απομείωση δεν σημαίνει αυτό ότι δεν θα υπάρξει ε, στρατιωτική ε, αντίσταση. Υπάρχει συρρήκνωση. Υπάρχουν κάποιες ενδείξεις ότι ένας μεγαλύτερος αριθμός ατόμων που διασυνδέονται με την Αρσαμπάμπ είναι άτομα και μικρότερες ομάδες που δείχνουν ότι έχουν την πρόθεση να αποσυνδεθούν από την Al-Shabaab στο μέτρο που υπάρχουν τώρα σοβαρότερες συζητήσεις για το πώς θα πρέπει να αντιμετωπιστεί αυτή η προσπάθεια αυτών των ατόμων να αποσυνδεθούν από την Al-Shabaab. Λοιπόν, στο ένα επίπεδο δεν θα πρέπει να υποθέσει κανείς ότι όταν λέω ότι υπάρχει απομείωση, συρρήκνωση της al ότι υπάρχει μια τακτική μετάθεση, ο αριθμός τους μειώνεται, αλλά ο σκληρός πυρήνας υφίσταται και με ασυμμετρικές μεθόδους ε, μπορούν να είναι πάρα πολύ επικίνδυνοι και ε, ε, πολύ ε, σκληροί αντίπαλοι. Τώρα, σε σχέση με αυτές τις συζητήσεις ή επαφές με την ε, Θα πρέπει να δούμε ότι πρέπει να τηρηθεί ε, εχεμήθεια και να είμαστε προσεκτικοί. Οποιοςδήποτε επιλέγει και επιδεικτικά αποσύρεται από την άσκηση βίας θα πρέπει να μπορεί να είναι ένα άτομο με το οποίο μπορούμε να έχουμε επαφή και να έχουμε επαφή με αυτό ώστε να μπορέσει να συνεχιστεί αυτή η θετική προσέγγιση. Έτσι θα πρέπει να ξεκινήσουμε σε περίπτωση που υπάρξει μια τέτοια κίνηση και τέτοια άτομα απεμπολίσουν τη βία και θελήσουν να επανενταχθούν στην κοινωνία, να μπορέσουν να συζητηθούν θέματα αμνηστίας, αμνίστευσης για τέτοιους ανθρώπους και έτσι να τους προσεγγίσουμε. Όπως είπα και προηγούμενα, υπάρχουν πολλοί οι οποίοι εμπλέκονται ε, στο επίπεδο αυτό. Οι Σομαλοί γνωρίζουν ο ένας τον άλλον σε σχέση με τις ε, επαφές τους για το τι κάνει ο ένας ή ο άλλος. Αυτό δεν σημαίνει ότι αν ο ένας βρίσκεται στη μία, στο ένα επίπεδο ή στο άλλο δεν έχουν επαφή και δεν γνωρίζουν ο ένας για τον άλλον. Αυτό είναι ένα από τα ξεχωριστά στοιχεία της Σομαλία. Δεν μας ε, εκπλήσει αυτό. Υπάρχουν και άλλοι εμπλεκόμενοι όμως στη Σομαλία. Δεν είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση και μια ε, ομάδα λευκών οι οποίοι θα αισθανόντουσαν καλά για την βοήθεια που θα παρεχόταν στην Σομαλία. Υπάρχουν κοινωνίες και στρώματα ολόκληρα που ε, είχαν και έχουν επαφές με τους Σομαλούς και θα εξακολουθούν να τις έχουν όταν εμείς ε, θα έχουμε αποχωρήσει. Ο, κόσμο, αραβικός κόσμος έχουν τέτοιες σχέσεις λοιπόν. Πρέπει να ακούσουμε πολύ προσεκτικά ποιες είναι οι δικές τους προτάσεις, οι δικές τους ιδέες, προτάσεις και αυτά τα οποία θα ήθελαν να προαγάγουν. Υπό αυτό το πρίσμα πρέπει να το προσεγγίσουμε ως Ευρώπη αντιμετωπίζοντας το θέμα της Σομαλίας. Το θέμα της επαρκούς χρηματοδότησης με κονδύλια να αποσαφηνίσω αυτό το οποίο ήθελα να πω. Πιστεύω ότι υπάρχουν αρκετά κονδύλια, επαρκή κονδύλια που δεσμεύονται για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη για τη Σομαλία και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από πολλές άλλες χώρες και θεσμικά όργανα που και αν υπό τις σημερινές προϋποθέσεις και όρους. Θα έπρεπε να τα εξετάσουμε προσεκτικά και να πούμε ορίστε αυτά είναι τα σχέδια, αυτά είναι τα κονδύλια αλλά μια και υπάρχει μια μετάθεση κέντρου βάρους ε, ή στόχων θα πρέπει να δούμε και την αναμετάθεση, αναδιαμόρφωση και όχι μόνο ε, ε, εν μέρη αλλά συνολικά θα μπορούσαμε να είχαμε ένα πολύ αποφασιστικό αποτέλεσμα με μια τέτοια σωστή δράση λαμβάνοντας υπόψη τις πολιτικές πραγματικότητες. Η πολιτική δράση στην πολιτική πραγματικότητα πρέπει να έχει κίνητρα. Κίνητρα που θα προσφέρονται στους, ε, στα άτομα στις, ε, σε μια κοινωνία. Αυτό είναι που πρέπει να λάβουμε υπόψη. Να θέλουμε να στεφτεί με επιτυχία το εγχείρημά μας να διασφαλίσουμε την παροχή ασφάλειας, να διασφαλιστεί ένα πλαίσιο ασφάλειας για τους Σομαλούς και τη Σομαλία. Για τη Σομάλι, την, το Σομάλι Λάντα σημειώθηκε και ε, λαμβάνεται υπόψη και νομίζω ότι και εσείς κατανοείτε κατανοείτε αυτό που θέλω να πω. Πρέπει να είναι σαφές. Το βλέπουμε αυτό και όταν το βλέπουμε αυτό παντού είναι σημαντικό να το λάβουμε υπόψη. Θα προτιμούσα η Αφρικανική Ένωση, τα κράτη της Αφρικανικής Ένωσης ε, να μπορέσουν ε, να δραστηριοποιηθούν επαρκώς. Ένα πράγμα όμως πρέπει να μας απασχολήσει η Σομάλιλαντ και η ηγεσία της πρέπει να το λάβει υπόψη. Οτιδήποτε θέλουν να πετύχουν οι ίδιοι πρέπει να διαρωτηθούν ποιες θα είναι οι επιπτώσεις και το τι θα συνεπάγεται το μέτρο και η φύση των δράσεών τους σε μια τέτοια πολύ ευαίσθητη περιοχή. Ποιες επιπτώσεις θα είχαν αυτές οι δράσεις. Είναι στα προς το συμφέρον της Σομάλιλαντ θα έλεγα να συνεισφέρει με κάθε εφικτό δυνατό τρόπο ώστε να συνεισφέρει ώστε η ίδια η ε, Σομαλία να είναι ε, δυνατό να επιβιώσει και να ε, αναπτυχθεί. Απλά και μόνο αναφέρομαι κάνουμε σε σχέση με εκείνα τα οποία ε, θα ήθελαν να αναλάβουν ως ε, ε, πολιτική δράση και πρωτοβουλίες. Πρέπει να το δουν αυτό μέσα στην πολιτική πραγματικότητα που είναι ιδιαίτερα ευάλωτη και ευαίσθητη για την συνεισφορά με ιδέες ή προτάσεις για το πώς θα μπορούσε να επιληθεί ένα πρόβλημα που είναι περιφερειακό πρόβλημα και έχει επιπτώσει στην ευρύτερη περιφέρεια και όχι μόνο σε μια περιοχή ή χώρα. Αν θέλουν λοιπόν να επιτύχουν κάτι πρέπει να δούμε ποιες θα είναι οι επιπτώσεις στο σύνολο της περιφέρειας αυτής. Νομίζω κάλυψα τις περισσότερες παρεμβάσεις για τα πλοία. Υπήρξε η ερώτηση του τι έκαναν οι Αμερικανοί υπό το φως αυτό. Δεν έχω εγώ τα εχέγγια να απαντήσω σε αυτή την ε, ερώτησή σας και δεν μπορώ να δώσω απάντηση. Ευχαριστώ. Μια αντίστοιχη παρατήρηση που έγινε και για τη Ρωσία προηγουμένως. Αυτό το οποίο μπορώ να πω είναι ότι συνεργαζόμαστε στενά με τους Αμερικανούς σε επίπεδο θαλάσσια στρατιωτική παρουσίας συμμετέχουν οι Αμερικανοί είτε δίδοντας σκάφη στο ΝΑΤΟ είτε προσφέροντας τι ε, δικές τους μονάδες. Συνεργαζόμαστε μαζί τους ε, σε καθημερινή βάση. Την προηγούμενη εβδομάδα ήμουνα στο Μπαχρέιν και συζητούσα μετά της πειρατεία ε, με τον αρχηγό της μαχικής δύναμης εκεί. Δεν γίνεται λοιπόν κατα... περιστασιακά η συνεργασία, αλλά λειτουργούν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες και σε καμία περίπτωση δεν επαληθεύω αυτό το οποίο είπατε προηγουμένως. Μια συμπληρωματική ερώτηση. Ο κύριος Κυριλόφ, συμπληρωματική ερώτηση. Η ερώτησή μου θα τη με απλό τρόπο. Υπάρχει μία κάποια, θα έλεγα, τάση μείωσης επιθέσεων εναντίον των σκαφών με αμερικανική σημαία. Μετά από την τελευταίες ενέργειες των Αμερικανών. Μήπως θα πρέπει εν πάση περιπτώσει να γίνετε πιο άγριοι ε, για να σας πάρουν σοβαρά. Κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι έχουμε κάποιες αποδείξεις που στηρίζουν τον ισχυρισμό σας. Υπάρχουν ε, κάποιες ε, ενδείξεις σύμφωνα με την δράση σκληρή την οποία ανέλαβαν οι Ινδοί απέναντι στους πειρατές κοντά στις ακτές τους και το ότι δεν είδαμε πειρατές να δραστηριοποιούνται σε αυτή την περιοχή ε, φέτος, αυτό είναι σαφές. Από την άλλη δεν τους είδαμε επίσης να λειτουργούν ούτε και σε, ε, στην περιοχή της Αραβικής θάλασσας. Υπάρχουν λοιπόν κάποιες ενδείξεις οι οποίες θα μπορούσαν να επινευτούν ότι οι πειρατές αντιμετωπίζουν διαφορετικές χώρες με διαφορετικό τρόπο και θα έλεγα ότι οι πείρατες ε, δεν είναι απόλυτα ενημερωμένοι ε, και δεν μπορούν να γνωρίζουν ε, τι είναι τα σκάφη τα οποία θα έλεγα είναι αυτά τα οποία, στα οποία επιτίθενται. Επιτέθησαν σε δύο στρατιωτικά σκάφη χωρίς να το γνωρίζουν προφανώς και γι' αυτό και φυσικά ιτήθηκαν και συνελήφθηκαν. Δεν νομίζω λοιπόν ότι έχουν αυτή τη διακριτική ευχέρεια να γνωρίζουν τους στόχους τους οποίους επιτίθενται. Ο κύριος Ρόντος, ένα επιπλέον σημείο. Και μετά Γκάλερ και Λόιζινγκ. Ένα πολύ σημαντικό θέμα το οποίο τέθηκε για το εάν η ενιοποίηση, η ενοποίηση όλων των στρατιωτικών δυνάμεων υπό την ηγεσία των Ηνωμένων Εθνών θα ήταν χρήσιμη. δεν ξέρω αν μπορεί να συγκρίνει κανείς σε διαφορετικές καταστάσεις. Υπάρχει πράγματι μία πολλαπλότητα, αν θέλετε, ευθυνών. Στη Σομαλία όμως. Ο ειδικό αντιπρόσωπος των Ηνωμένων Εθνών είναι υπεύθυνο για τις πολιτικές διαδικασίες. Από ό,τι γνωρίζω δεν ελέγχει τις στρατιωτικές ενέργειες τις οποίες είναι υπεύθυνη η Αφρικανική Ένωση και δεν ελέγχει ο εκπρόσωπος του ΟΗΕ ε, τα αναπτυξιακά προγράμματα και τις αναπτυξιακές πιστώσεις. Αυτό σας το λέω για να κατανοήσετε πώς έχει η κατάσταση και πώς λειτουργεί σε επίπεδο Ηνωμένων Εθνών. Γιατί όπως είπα ότι αυτά ε, εντάσσονται στα πλαίσια της εντολής του Συμβουλίου Ασφαλείας. Νομίζω λοιπόν ότι έχουμε φτάσει σε μια φάση πλέον και τίθεται το θέμα για μια ολοκληρωμένη αντιμετώπιση. Ε, επιθυμούμε εμείς να εμπλακούμε σε μια σε εισαγωγικά συζήτηση για το ποιος έχει τι, τι μπορεί να κάνει και τι μπορεί και πράγματι να προσφέρει. Ή μήπω θα πρέπει να συγκεντρώσουμε την προσοχή μας σε αυτά τα οποία μπορούμε να κάνουμε με ολοκληρωμένο τρόπο με τις δυνάμεις που έχουμε στη διάθεσή μας. Εγώ προτιμώ αυτήν την στάση, αλλά παρόλα αυτά ίσως να έρθει κάποια στιγμή ή στιγμή όπου θα φανεί ότι δεν μπορούμε εμείς να θυσιάσουμε τις θυσίες που έχουμε, τις προσπάθειες που έχουμε κάνει στη Σομαλία στα πλαίσια μιας ευρύτερης προσπάθειας βελτίωσης των αρχών λειτουργίας της παρέμβασής μας. Γκάλερα. Ήθελα να ε, τελειώσω με μια θετική παρατήρηση. Ε, αλλά σε ελέγξουμε ποια ήταν τα τελευταία νέα του BBC για την Σομαλία. Ήταν εντυπωσιακό το ότι ακούσαμε ότι ξανά άνοιξε το Εθνικό Θέατρο της Σομαλίας ε, και ε, υπήρξε μια παράσταση ενός ε, musical μετά από 20 χρόνια. Ε, βεβαίως αυτό είναι κάτι ευχάριστο και μας δείχνει ότι τα πράγματα πηγαίνουν προς τη σωστή κατεύθυνση όταν οι άνθρωποι έχουν τη δυνατότητα να ξανανοίξουν το Εθνικό Θέατρο και αυτό σχετίζεται με τα όσα είπατε για την ζωή, τον παλμό που υπάρχει στην πόλη. Άρα λοιπόν κάπου αισθάνομαι ότι επιβεβαιώνομαι από τα ίδια τα νέα της ειδήσει. Γιατί ήταν πρώτη φορά μετά πολύ καιρό που είχαμε μια τόσο ευχάριστη είδηση. Η κυρία Λούζινγκ έχει το λόγο. Θα ήθελα να αναφερθώ σε αυτό το οποίο μόλις είπε ο κύριος Στένοκ. Ε, πρόκειται για μια μικρή παρανόηση. Εγώ δεν μίλησα με γενικού όρους, αλλά είπα ότι θα πρέπει να υπάρχουν διαφορετικές συνθήκες κράτησης για ανήλικους και ενηλίκους. Ε, ε, και ε, αν δούμε τι γίνεται στο Αμβούργο και θεωρώ ότι είναι μια ρατσιστική πρακτική και δεν είναι συμβατή με τους κανόνες ενός κράτους δικαίου και νομίζω ότι τα πράγματα θα είναι καθόλου διαφορετικά και στην ε, Μεγάλη Βρετανία. Δεν είναι δυνατόν να υπάρξουν ίδιες, δεν θα υπάρχουν και εκεί ίδιες φυλακές για ενηλίκους, για μεγάλους άνδρες όπως για τους ε, νεαρούς, τους ανηλίκους. Δεν ξέρω, θέλετε να προσθέσετε κάτι εν κατακλείδη. Εάν όχι, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για την ε, παρουσία σας, ιδιαίτερα τον Άλεξ που έκανε ένα τόσο μεγάλο ταξίδι για να μας συναντήσει. Νομίζω ήταν μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συνεδρίαση και οι προσπάθειες που γίνονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτή την περιοχή του κόσμου ε, δείχνουν ε, πλήρως τις, τους ολόδοξους που έχει θέσει η συνθήκη της Λισαβόνα σε θέματα ε, ασφάλειας, ε, πολιτικής ασφαλείας. Και νομίζω ότι οι προσπάθειες αυτές ε, θα πρέπει να συνεχίσουν σε συντονισμό με όλους τους άλλους φορείς και όλες τις άλλες χώρες μέλη που ενδιαφέρονται για τις εξελίξεις σε αυτή την περιοχή ε, θεωρώ ότι έχει νόημα να συνεχίσουμε μια σβάθος συζήτηση μαζί σας γιατί η περιοχή αυτή στο κέρας της Αφρικής μαζί με το Σαχέλ που είναι μια περιοχή της Αφρικής όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση αναλαμβάνει όλο και περισσότερο ενεργό δράση είναι μια πολύ σημαντική περιοχή για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είσαι σε αυτή την ε, επιτροπή ε, γιατί θα πρέπει να είμαστε και εμείς ενήμεροι για τις εξελίξεις. Είδατε ότι ορισμένοι από εμά ε, ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για τα τεκτενόμενα σε αυτή την περιοχή. Σας ευχαριστούμε πολύ. Θα επανέλθουμε σήμερα το μεσημέρι με μια ενημέρωση όσον αφορά τις επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ ε, στη Λιβύη τον περασμένο χρόνο με τον εκπρόσωπο του ΝΑΤΟ εδώ στις ε, Βρυξέλλες.